So, Kolleginnen und Kollegen, ich würde sagen, dass wir Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ. Και θα ξεκινήσουμε με το σημείο 26 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε ένα προσκεκλημένο εδώ σήμερα, τον ε, Δόκτωρο Φρόσκ, και θα μας κάνει σήμερα μία παρουσίαση σχετικά με την ειδική έκθεση ε, σχετικά με την ε, διαχείριση των ε, συγκρούσεων συμφέροντος σε κάποιους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για να κάνετε την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θα μιλήσω αγγλικά, μου επιτρέπετε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη πρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι σήμερα ενώπιόν σας και ε, σας ενδιαφέρει να παρουσιάσω την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφέροντος σε συγκεκριμένων χρονών που δημοσιεύθηκε στο Δεκέμβρη. Θα ήθελα να πω το θέμα της σύγκρουση ε, συμφερόντων είναι ένα ζήτημα το οποίο ξεκίνησε στη δική σας επιτροπή ήδη το 2009. Άρα μπορώ εν μέρη να αφήσω κάποια σημεία τη παρουσίασή μου και να μην εξηγήσω γιατί είναι τόσο σημαντικό θέμα η σύγκρουση συμφερόντων. Θα ξεκινήσω λέγοντας γιατί επέλεξε το ελεκτικό συνεδρίο αυτό το θέμα και πώς επέλεξε τους οργανισμούς για τον έλεγχο. Θα θυμάστε ίσως ότι τον, την άνεξη του 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ζήτησε έναν έλεγχο με περιστατωμένη ανάλυση τη προσέγγιση που ακολουθούν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί για τη διαχείριση καταστάσεων όπου υπάρχει ε, ενδεχόμενο σύγκρουση συμφερόντων. Είδαμε μια σειρά φερόμενων υποθέσεων που θα μπορούσαν να ταχθούν στην κατηγορία σύγκρουση συμφερόντων και αφορούν συγκεκριμένου ευρωπαϊκού οργανισμού που ε, συχνά καταγγέλνουν στον τύπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη διάθεσή τη μια ε, ευρεία γκάμα οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με ακόμη ευρύτερη γάμα θεμάτων. Και μάλιστα πολλοί τέτοιοι οργανισμοί λαμβάνουν αποφάσει για θέματα ασφάλεια, υγεία των εργαζομένων, των καταναλωτών, ε, ασφάλεια τροφίμων, μεταφορέ κτλ. Η αξιολόγηση του ε, Ελεκτικού Συνεδρίου αξιολόγησε πολιτικέ και διαδικασίε για τη διαχείριση σύγκρουση συμφερόντων σε τέσσερι επιλεγμένε ε, υπηρεσίε. Πρώτα απ' όλα την ασφάλεια της Αεροπλογίας, την υπηρεσία για τα χημικά, την ε, ΕΦΣΑ και την, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων με στόχο να απαντήσουμε στα εξή ερωτήματα. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν καταφέρει αποτελεσματικά να διαχειριστούν περιπτώσει συγκρούση ε, συμφέροντο. Και προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα σχετικά. Πρώτον, υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίε για να διαχειριστούν συγκρούσεις συμφέροντος. Και το δεύτερο ερώτημα, οι επιλεγμένοι οργανισμοί έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά τις πολιτικές για τη διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων συγκρούσεων συμφέροντος. Βεβαίω, ότι και σε ειδικέ εκθέσει προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και συστάσει για τα ίδια σημεία. Για να γίνει αυτό ο έλεγχο, έπρεπε να ορίσουμε κάποιε παραμέτρου πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, εν τη απουσία ενός ορισμού της έννοιας σύγκρουση συμφερόντων, ήταν πολύ χρήσιμος ορισμός των κατευθύνων γραμμών του ΟΣΑ. Δεύτερον, έπρεπε να ορίσουμε ένα πλαίσιο αναφοράς με ελάχιστες απαιτήσει σχετικά με την εξαρτησία και τη διαφάνεια των βασικών παικτών που συμμετέχουν στις διάφορες διαδικασίες των οργανισμών. Επίσης, κρίθηκε αναγκαίο να αποταθούμε και πάλι στις κατευθύνες γραμμές του ΩΣΑ με διεθνή benchmarks που αφορούν ακριβώς την πολιτική και την αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων συμφέροντος. Τώρα θα πάω ε, στα συμπεράσματα των ε, αρμόδιων του Ελεκτικού Συνεδρίου. Εστιάσαμε στις διαδικασίες και τις πολιτικές και την διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων συγκρούσεων συμφέροντος Ανέφερα πριν τους τέσσερις επιλεγμένους οργανισμούς. Το πρώτο πόρισμα ήταν ότι δεν υπάρχει ένα εμπεριστατωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο που να αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων ώστε να καταλήξουμε σε συγκρίσιμα ε, προϋποθέσεις σχετικά με τη διαφάνεια και να αφορά όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους πορίσματα, η εικόνα είναι μεικτή. Αλλά να ξεκινήσουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα καταλήξουμε συμπέρασμα ότι οι επιλεγμένοι οργανισμοί ε, αντιμετώπισαν επαρκώς τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφέροντος. Πρέπει να πω όμως ότι ε, εντοπίστηκαν κάποια επίπεδα ελλημάτων ε, και προβλημάτων στους οργανισμούς που διέφεραν σε επίπεδο και εύρος. Αυτό φαίνεται στην, στον πίνακα μετά την παράγραφο 89, όπως και στα παραρτήματα 3 και 4. Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Συνέδριο κατέληξε στα εξή. Από του επιλεγμένου οργανισμού, ο Οργανισμό Φαρμάκων και ο Οργανισμό ε, Ασφάλεια Τροφίμων έχουν τι πλέον εξελιγμένε πολιτικέ και διαδικασίε αντιμετώπιση ε, του φαινομένου. Ο Χημικό Οργανισμό είχε έναν ανεπαρκή και όχι απόλυτα ακριβή διαδικασία, ενώ ο ε, Οργανισμό για την Ασφάλεια Τροπλοή δεν είχε καμία τέτοια πολιτική. Γενικώ πώς οι επιλεγμένοι οργανισμοί δεν έχουν τους κατάλληλε τις πολιτικές και διαδικασίες για να αντιμετωπίσουν μία ειδική περίπτωση ε, ε, για να αντιμετωπίσουν ε, την κατάσταση. Γι' αυτό σε διαφορετικές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν επιρογνώμονες και μέλη πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου ελεκτικού οργάνου. Έπειτα δεν υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις αφήσει δήλωση ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερομένους και δεν υπήρχαν τα κατάλληλα κριτήρια, όπως είπαμε, τα οποία να εφαρμόζονται συνεπώς πάντοτε. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, την εφαρμογή της πολιτικής και των διαχειρήσεων των διαδικασιών συγγνώμη, στον οργανισμό χημικών, εκεί και εντοπίσαμε ελλείμματα. Σε ό,τι αφορά την ε, διαφάνεια και την τελική δήλωση ε, συμφερόντων καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όλοι οι επιλεγμένοι οργανισμοί εκτός από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας στην Αεροπλοεία ε, τα πράγματα ήταν ικανοποιητικά. Στον τελευταίο οργανισμό υπάρχει λιγότερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη δήλωση συμφερόντων ε, μεταξύ των επιστημονικών φορέων που απαρτίζουν ε, τα κατάλληλα όργανα. Από την πλευρά μας εξετάσαμε και την εκπαίδευση για την αντιμετώπιση ε, του φαινομένου και ότι θα έπρεπε να υπάρχει παντού. Όμω, στον Οργανισμό Χημικών και στον Οργανισμό Ασφάλεια στην Αεροπλοεία εντοπίσαμε και πάλι ελλείμματα στην εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό Ασφάλεια Αεροπλοεία, υπήρχαν προβλήματα στην εκπαίδευση όπως είπαμε και στον οργανισμό για τις χημικές ουσίες. Επίσης εξετάσαμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουν επιλεγμένοι οργανισμοί όταν οι υπάλληλοι και εμπειρογνώμονες εγκαταλείπουν τους οργανισμούς για να εργαστούν στο ιδιωτικό τομέα. Εκεί εντοπίσαμε μια σειρά ελλημάτων ως προς τα εξή, συγκεκριμένα. Έλλειψη διατάξεων για να αντιμετωπίσουν κινδύνους που συνδέονται με τις, ε, την εργασία που αναπτύσσουν ε, όταν εγκαταλείπουν τον οργανισμό. Έπειτα, από ε, ε, έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων ως προς τον ορισμό του τι είναι σύγκρουση συμφέροντων και τρίτον διαπραγμάτευση για μελλοντική απασχόληση που δεν καλύπτεται από τις εφιστάμενες πολιτικές διαδικασίε των οργανισμών. Τέλος, καταλήξαμε ότι μόνο ο Ευρωπαϊκό Οργανισμός Φαρμάκων έχει μια πολιτική για τι προσκλήσει και τα δώρα για όλο τον οργανισμό για να αντιμετωπίσουμε τι δυναμίε, καταλήξαμε σε μια σειρά συστάσεων που βλέπετε λεπτομερώ στην έκθεση και ακολουθούν τη λογική των συμπερασμάτων μας. Συστήνουμε για παράδειγμα ότι όλοι οι επιλεγμένοι οργανισμοί θα πρέπει να ορίσουν ή να αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες για τη σύγκρουση συμφερόντων, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά συγκεκριμένους κινδύνους. Ε, οι επιλεγμένοι οργανισμοί θα πρέπει να περνούν ή οι υπάλληλοι των οργανισμών να περνούν screening πριν α, ε, α, ε, λάβουν τη θέση και προσληφθούν. Και αυτό πρέπει να αφορά όλου του οργανισμού, όπω είπα. Οι επιλεγμένοι οργανισμοί θα πρέπει επίση να ορίσουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση τη δήλωση συμφερόντων και να εφαρμόζονται συστηματικά. Το ίδιο ισχύει και τη διαδικασία διαφάνειας που θα πρέπει να διέπει όλες τις εργασίες του οργανισμού για τον οργανισμό χημικών ουσιών συγκεκριμένα θα πρέπει να βελτιώσει καλύτερα την εφαρμογή των πολιτικών διαδικασιών για ε, τους υπαλλήλους ε, και το δευτεροβάθμιο όργανο. Θα μπορούσα να ε, προχωρήσω κυρίες και κύριοι αναφέροντας όλες τις συστάσεις του Ελληνικού Συνεδρίου αλλά θα μας πάρει χρόνο. Θα ήθελα να πω το εξή. Γιατί αναγνωρίζω ότι η ειδική επιτροπή δεν έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον για το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά πιο πολύ ενδιαφέρεται για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Υπ' αυτή την έννοια, να πω ότι μία από τις συστάσεις μας είναι η αριθμών 10 και 11. Ε, είναι δύο συστάσεις λοιπόν που λένε το εξή. Το τελικό συνέδριο θεωρεί ότι είναι μια καλή ιδέα ο Ευρωπαίος νομοθέτης σε διαβούλευση ίσως με άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ξεδάσει την περαιτέρω εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου με σκόπο τη διαχείριση των περιπτώσεων σύγκρουση συμφερόντων χρησιμοποιώντα βέλτιε πρακτικέ και ω σημείο αναφορά και τι τρεις γραμμέ του ΩΣΑ. Επίση, θα πρέπει να επισημάνουμε το εξή. Εμεί ολοκληρώσαμε τον έλεγχο τον Οκτώβριο του 2011 και άρα πρέπει να επισημάνουμε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη και πρόοδο είχαν οι οργανισμοί από τότε είναι κάτι που δεν έχει τύχει αξιολόγηση από εμά και δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την έκθεση. Κύριε Πρόεδρε, τελευταία τελευταία λίγα λόγια για το πώς έγινε αυτή η δουλειά από το ελεκτικό συνέδριο και θα θέλαμε να πούμε προκειμένο, ότι εξετάσαμε εντελεχώς περιπτώσεις και στους τέσσερις επιλεγέντες οργανισμούς με συναντήσει σε διάφορα επίπεδα. Εξετάσαμε εντελεχώς όλες τις ε, τις συνθήκες και καταλήξουμε συγκεκριμένες συστάσεις. Θεωρούμε λοιπόν τα συμπεράσματα, τα πορίσματα και οι συστάσεις μας έχουν ε, μια καλή βάση. Αυτά κύριε Πρόεδρε από πλευρά μου σχεδόν ολοκλήρωσα, αλλά θα ήθελα να πω σε αυτή τη φάση και κάτι ακόμα. Χωρίς την επικοδομητική στάση και των τεσσάρων επιλεγμένων οργανισμών κατά τη διαδικασία του ελέγχου, όπως και την τόσο καλά φωσιωμένη ομάδα ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου που δούλεψε για αυτό το θέμα, εγώ δεν θα είχα αυτή τη χαρά σήμερα να κάθομαι μαζί σας και να σας κάνω αυτή την παρουσίαση. Είμαι πραγματικά ευγνώμων ε, έναντι όλων αυτών και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις που μπορεί να έχετε επί του θέματος σε ευχαριστώ και πάλι για τη σημερινή πρόσκληση. Well, thank you very much, um, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και νομίζω ότι είναι πολύ καλό που επιτέλους έχουμε μια διαρθρωτική συζήτηση ε, πάνω στην ε, σύγκρουση συμφερόντων ε, που να μην βασίζεται απλά σε περιστατικά. Έχω κατάλογο ομιλητών Ε, μήπως υπάρχει κανένας άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Ο Μπαρτ Στάς πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσουμε το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη έκθεση και εγώ ανήκω στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και έτσι χαίρομαι που βλέπω αυτές τις ειδικές εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου είναι μία από τις εξαιρετικά ισχυρές, παρότι πάντα τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα των εκθέσεων ε, του ηλεκτρικού Συνεδρίου είναι πολύ καλά. Ε, την είχε προετοιμάσει αυτή την έκθεση και ο προκάτοχος, ε, το προηγούμενο μέλος δηλαδή του ηλεκτρικού συνεδρίου, θα ήθελα να, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Είπατε δικαίως ότι το εγχείρημα εδώ δεν είναι ένα εγχείρημα του παρελθόντος, αλλά του μέλλοντος και αυτό είναι η αρμοδιότητα και το καθήκον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ε, να έχει το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον. Το εγχείρημα για το, ε, του παρελθόντος συμβαίνει στην περίπτωση της απαλλαγής και πολύ ορθώς. Θα ήθελα όμω να θέσω ένα ερώτημα, όχι στο Ελεκτικό Συνέδριο, γιατί έχουν κάνει το έργο του, ε, αλλά προ την Επιτροπή. Στην εισαγωγή παραπέμψατε στι συστάσει 10 και 11. Ρητό ερώτημα λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σε ό,τι φορά την συμφωνία με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ε, διαχείριση των σημαντικών αυτών ε, διαφωνιών και συγκρούσεων. Το ερώτημα προς την Επιτροπή είναι το εξή. Είστε θετικά διακείμενε προ αυτό και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, πότε να περιμένουμε προτάσει. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όπως ε, ο συνάδελφος ε, τους προσκεκλημένους μας. Ήταν μια έκθεση που περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Είναι εξαιρετικά σημαντική για πολλούς ε, λόγους. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας το πιο σημαντικό στην Ένωσή μας είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών ε, στα, θεσμικά όργανα και στις αποφάσεις που λαμβάνουν. Στο πλαίσιο της σύγκρουσης συμφερόντων ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο επανέρχεται συνεχώς, ε, που υπονομεύει την εμπιστοσύνη που μπορούν να έχουν οι πολίτες μας στην ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται και στους λόγους για τους οποίους λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γι' αυτό ακριβώς και είναι τόσο σημαντική αυτή η έκθεση, γιατί ε, εξηγεί κάποια ζητήματα, αναλύει τα προβλήματα ε, που οδηγούν ε, σε κάποιε διορθώσει. Το πρόβλημα, Πρόεδρε, είναι ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Υπάρχουν και επιπτώσεις. Επιπτώσεις στις γνωμοδοτήσεις και ως εκ τούτου και στις αποφάσεις που όλοι μαζί λαμβάνουμε. Ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος χθε δημοσίευσε μια εξαιρετικά σημαντική έκθεση 800 σελίδων, ογκοδέστατη έκθεση και ε, ε, ομολογώ ότι δεν την έχω διαβάσει ολόκληρη ακόμα η οποία όμως δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες ανομαλίες ή κάποια λάθη σε ό,τι αφορά την, τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τις καθυστερήσεις. Αποφάσεις πολύ σημαντικές για την υγεία των πολιτών, ε, για το περιβάλλον και για ε, τα δημόσια οικονομικά. Καθυστερήσεις που οφείλονται στις ε, μελέτες και πραγματογνωμοσύνες και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι και αμφισβητήσιμες. Δεν θα πάω παραπέρα, όμως είναι κρίσιμη σημασία το θέμα. Δύο ερωτήματα λοιπόν. Ε, θα μπορούσε να λάβει και πάλι το ελληνικό συνέδριο και προς ε, σύντομα ε, το ίδιο ζήτημα για να δει πώς ε, ακριβώς έχει ανταποκριθεί ο κάθε οργανισμός στις επικρίσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεύτερο σημείο, όπως και ο συνάδελφος έθεσε προηγουμένως και απευθύνομαι προς την Επιτροπή, ε, θεωρείτε ότι θα έχετε μέχρι ε, το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας εντολή ούτω, ώστε να επεξεργαστείτε αυτό το θέμα επαρκώς ε, και ένα σημαντικό τμήμα των επικρίσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τον ρόλο των λόμπι, των ομάδων πίεσης, της αμφισβήτησης των γνωμοδοτήσεων των εμπειρογνωμόνων να μειωθεί χάρη σε αυστηρούς κανόνες και να ελέγξετε, το υπογραμμίζω αυτό, να ελέγξετε τις ε, δηλώσεις ε, συμφερόντων στη συνέχεια και τις ε, συγκρούσεις συμφερόντων στη συνέχεια που και θεωρώ ότι αν φτάσουμε μέχρι εκεί θα μπορούμε να διασφαλίσουμε σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνουμε και θα στηρίξουμε την, ε, θα αυξήσουμε μάλλον την εμπιστοσύνη των πολιτών μας ε, στους οργανισμούς μας, που είναι ε, θεμελιώδης σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κορίν Λεπάζ. Ε, να δώσω το λόγο στον καθηγητή για να απαντήσει σε, στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Παρακαλώ, το λόγο. Α, όχι, ένα λεπτό. Νόμιζα ότι είχατε πάρει το λόγο. Ζήτω ε, συγγνώμη, Πρόεδρε. Ε, δεν θα ήθελα να ξεχάσω τον εισηγητή. Παρακαλώ. Μπήκα στο τέλος ε, της, του καταλόγου γιατί ήμουνα στην θέση σας πριν από δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη να έχουμε ισχυρούς, ανεξάρτητους ε, και αξιόπιστου οργανισμού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να επιληθεί αυτό το πρόβλημα της σύγκρουση συμφερόντων. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν ε, ε, ε αποφάσεις ε, που ενδεχομένω να έχουν αμφισβήτηση σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Όμω, χαίρομαι που επιτέλους έχουμε μια τέτοια δομημένη ε, συζήτηση που δεν βασίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά όπως έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού είχαμε μια ακρόαση για την ε, απαλλαγή για το 2011 ε, ενός από τους οργανισμούς και για την συγκεκριμένη αυτή έκθεση. Το συζητήσαμε και σήμερα το πρωί. Έχω όμως ε, κάποιες παρατηρήσεις και ερωτήματα προς τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ απολύτω με την σύστασή σας να αναπτύξουμε τους, τις δικές μας κατευθυντήριες γραμμές, γιατί οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ δεν ε, επαρκούν, δεν ε, άπτονται όλων των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Για παράδειγμα, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν μόνο ε, τους εργαζομένους ε, των οργανισμών και όχι τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, που είναι ένα από τα πιο ακαθόδη ζητήματα για αυτούς τους οργανισμούς. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με αυτό. Και θα ήθελα να ρωτήσω και την Επιτροπή να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει ως προς αυτό. Ένα ερώτημα ε, προς το μέλος ε, του Ελεκτικού Συνοδριού ε, για το τι είδους συγκρούσεις συμφερόντων αντιμετωπίσατε και εξετάσατε μάλλον. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην έκθεση αλλά είναι σημαντικό, είναι η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ίδιου του οργανισμού και του Διοικητικού του Συμβουλίου με εκπροσώπου όλων των κρατομελών. Πολλέ φορές υπάρχουν και εθνικά συμφέροντα τα οποία αντικατοπτρίζονται στην ε, συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήδη αυτό μπορεί να αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων γιατί μπορεί να μην είναι προ το συμφέρον του οργανισμού. Υπάρχουν όμως και οργανισμοί όπου συμμετέχουν εθνικοί εκπρόσωποι εκ μέρου εθνικών οργανισμών και εκεί υπάρχει σαφής σύγκρουση συμφερόντων γιατί ε, αυτά τα εθνικά θεσμικά όργανα πολλές φορές ε, θεωρούνται άμεση ανταγωνιστές ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι γιατί δεν συμπεριλήφθη αυτό στην μελέτη σας. Ίσως θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να διαρευνήσετε στο μέλλον. Μπορούμε μετά να συζητήσουμε τον ίδιο το ρόλο των εθνικών εκπροσώπων σε αυτά τα διοικητικά συμβούλια. Γιατί νομίζω ότι ένας ε, ανεξάρτητος και αξιόπιστος οργανισμός δεν θα πρέπει ε, να έχει ε, στις γραμμές του εθνικούς εκπροσώπους που ουσιαστικά υπερασπίζονται εθνικά συμφέροντα. Τέλος, Πρόεδρε, σήμερα το πρωί ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΦΣΑ έκανε μια δήλωση ότι θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στην εσωτερική πραγματογνωμοσύνη, δηλαδή να μην απευθύνονται σε εξωτερικούς ε, εμπειρογνώμονες από πανεπιστήμια ε, και ούτω καθεξής, αλλά μέσα στον οργανισμό, ιδίως για τα ε, λεπτά και ευαίσθητα ζητήματα, όπως οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, όπως συμβαίνει και στι ε, στις ΕΙΠΑ όπου έχουμε τον Οργανισμό Περιβαλλοντικής Προστασίας. Το ερώτημά μου προς την Επιτροπή και προς το Ελληνικό Συνέδριο θα ήταν αυτό μια καλύτερη λύση που θα διασφαλίζει την απόλυτη ανεξαρτησία. Θα ήταν αυτός ο καλύτερος τρόπος για να επιληθεί η σύγκρουση συμφερόντων και είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το κόστος γιατί θα είναι πολύ πιο ακριβό από το υφιστάμενο σύστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ εξετάζουμε ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για τη σύγκρουση των συμφερόντων. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι δηλαδή πρέπει πράγματι να υπάρχει έλεγχος. Όμως ε, όταν υπάρχει έλεγχος αλλά δεν υπάρχει κύρωση τότε αυτό δεν έχει νόημα. υπάρχει εδώ πέρα η πολιτική των κυρώσεων όμως ουσιαστικά πρέπει να έχουμε απτές κυρώσεις κάποια στιγμή και με όλες τις συγκρούσει συμφερόντων που είχαμε στου οργανισμούς ε, πολύ συχνά υπόθηκε ναι αλλά τα κράτη-μέλη είναι αυτά που διαλέγουν τους εμπειρογνώμονες. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σε επίπεδο οργανισμού υπάρχει ένα κύτταρο που διασφαλίζει ότι αν ο πυρογνώμονα ε, που αποστέλλεται από ένα κράτο μέλο δεν ε, ανταποκρίνει τι υποχρεώσει του, τότε δεν επιλέγεται και τους παρέχουμε άλλες, άλλους εμπειρογνώμονες που δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα, κάτι το οποίο εμένα με εξέπληξε που αφορά τη διοίκηση. Για παράδειγμα, Γενική Διεύθυνση ε, ΣΑΝΚΟ ή Ανταγωνισμού, ή Ενέργειας. Γνωρίζετε ότι δεν τους ζητάμε δήλωση συμφερόντων. Και αυτό είναι μια δυσλειτουργία πώς είναι δυνατόν οι γενικοί διευθυντές να μην οφείλουν να υποβάλουν ε, δήλωση ε, συμφερόντων ενώ υπάρχει δρακόντια πειθαρχία και δρακόντια μέτρα ε, στους υπολείπους. Φανταστείτε ότι η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ επιβάλλει κυρώσει ε, ε, στη βιομηχανία, ενώ ήδη δεν έχουν καμία υποχρέωση. Υπάρχει λοιπόν ε, μια τέτοια ανισορροπία. Και ένα τρίτο στοιχείο που με έχει εκπλήξει είναι ότι και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα, όταν ορίσαμε την Ισελ επικεφαλής ε, της ε, Επιτροπής Δεντολογίας ε, που εξετάζει τις δαπάνες των επιτρόπων μετά την αποχώρησή τους. Εκείνη Εκείνος συγγνώμη, ήταν μέλος των υπηρεσιών της Επιτροπής και τώρα βρίσκεται στο Υπουργικό Συμβουλίο του Διοικητικό Συμβούλιο της Φίλιπ Μόρι, του Κολοσσού της Καπνοβιομηχανίας. Πώ είναι δυνατόν λοιπόν να εμπιστευόμαστε ένα τέτοιο έργο σε κάποιον που ε, βρίσκεται βυθισμένο μέσα στη σύγκρουση συμφερόντων. Αν θέλουμε να το κάνουμε λοιπόν αυτό σε επίπεδο οργανισμών, πρέπει να το κάνουμε σε όλα τα επίπεδα, και με έλεγχο και με κυρώσει, για να αυξηθεί και αξιοπιστεί απέναντι στους ευρωπαίου πολίτε. Gut, jetzt erhält dann abschließend... Το λόγο έχει ο δόκτωρο για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Στές για τα ευγενή του λόγια, για τη δουλειά που κάναμε. Πράγματι, όλη αυτή η δουλειά ξεκίνησε από τον προκάτοχό μου, από τον κύριο Σίμα τον Ιρλανδό συναδελφό. Εγώ ε, συνέχισα αυτό το έργο από πέρυσι. Σε όσα είπε τώρα η κυρία Λαπάζ, αν κατάλαβα καλά, ρωτήσατε τι συνέχεια προβλέπει να δώσει το ηλεκτρικό συνέδριο στο μέλλον. Όπως συμβαίνει με κάθε έκθεση, το ηλεκτρικό συνέδριο θα εξετάσει εν ευθέτω χρόνο Ποιο είναι ο κατάλληλο τρόπο να δώσει συνέχεια στο θέμα. Σε αυτή την περίπτωση, Ίσως σας ενδιαφέρει να σας πω ότι η Κομισιόν στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς προετοίμασε ένα roadmap για την ε, συνέχεια στην παρακολούθηση της κοινή προσέγγισης στους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Και μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται είναι το, η σύγκρουση συμφερόντων. Και αν δεν κάνω το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε είναι τα τέλη αυτής της χρονιάς. Τι θέλω να πω. Αυτό που είναι σημαντικό για μας και ελπίζω και για σας, πω όλα, θα ξεκινήσουμε μία πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τις πολιτικές διαδικασίες για τη σύγκρουση συμφερόντων. Και μετά ελπίζουμε να υπάρχει ευκαιρία να εφαρμοστούν. Άρα, καλό θα είναι να επανέλθουμε να δούμε τι συμβαίνει. Να δούμε αν πραγματικά υπάρξει, υπάρχει βελτίωση ή όχι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα υπάρξει σίγουρα follow-up, θα υπάρχει συνέχεια από εμά. Αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή. Σίγουρα δεν είναι κάτι που γίνεται μια φορά και θα το ξεχάσουμε. Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα του κ. Γκεμπράντη, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Στην αρχή της έκθεσης έχουμε μια σειρά σημείων που θεωρούμε ότι είναι οι εγγενείς ε, κίνδυνοι μέσα σε κάθε οργανισμό και από όπου ελοχεύει ο κίνδυνος της σύγκρουσης συμφερόντων. Οπότε σίγουρα δεν είναι κάτι που μας διέφυγε. Εγώ πιστεύω ότι προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλους τους κύριους ε, κινδύνους σύγκρουση συμφερόντων ή τουλάχιστον πιο πολλούς. Έπειτα, αν κατάλαβα καλά το insourcing που ετέθηκε σήμερα το πρωί από ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Δίκιο έχετε. Θα είναι πιο δεπανηρό άμα γίνει αυτό. Αυτό όμως θα επιφέρει την κατάλληλη ισορροπία και κατά πόσο θα υπάρχει μια ικανοποιητική πόσο θέλω. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, δεν είμαι ειδικό. Σίγουρα πρέπει να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία. Κατά πόσο δηλαδή οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται όσο γίνονται αυτή τη στιγμή από ε, το ελεκτικό συνέδριο και μόνο, δηλαδή να γίνεται με το insourcing, ή θα πρέπει να το κάνουμε όπως γίνεται σήμερα, με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς. Κατανοώ μεν το πρόβλημα που επισημαίνεται, αλλά δεν έχω μια εύκολη λύση να την προτείνω. Το σχόλιο της κυρίας Ριβαζή. Πράγματι, δίκιο έχετε. Στις συστάσεις μας είμαστε πολύ ε, προσεκτικοί. όταν λέμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ε, ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Εσείς δίκιο έχετε. Αυτό δεν πρέπει να αφορά μόνο στους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα πρέπει να αφορά και άλλους φορείς όπως ε, τις κοινές, ε, από τις κοινοπραξίες. Το θέμα είναι σε τι επίπεδο θα πρέπει να έρθει αυτό το κοινό και τι θα πρέπει να αφαιθεί στην ευθύνη του καθενός και σε επίπεδο οργανισμών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι απάντησε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις και για την παρουσίασή σας εδώ σήμερα. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη ε, να διορθωθούν κάποια πράγματα και σε άλλα θεσμικά όργανα θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Είναι μόνιμο καθήκον να επιδιώκουμε συνέχεια βελτίωση της κατάστασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φτάνουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, που είναι η οδηγία για το μέλη. Ε, μπορώ να πάρω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ε, ναι, αλλά έθεσα μια ερώτηση και προς την Επιτροπή. Δεν ξέρω αν είναι παρούσα η Επιτροπή. Η κυρία Λεπάζ αναφέρθηκε στα συμπεράσματα 10 και 11 ε, που τίθεται προς την Επιτροπή επίσης. Αν είναι παρούσα η Επιτροπή θα ήθελα να απαντήσει. αν όχι, θα, νομίζω θα ήταν χρήσιμο να λάβουμε γραπτή απάντηση. Είναι η Κομισιόν σε θέση να απαντήσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, πράγματι είμαι εκπρόσωπο ε, τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. επομένω ε, δεν μπορώ να εκπροσωπήσω όλε τι ε, γενικέ διευθύνσει που εξετάζονται εδώ, αλλά μπορώ να απαντήσω στα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Υγεία Καταναλωτών. Και ιδίω στα όσα αναφέρθηκαν για τη Γενική Διευθύντρια και η πρόταση που κατατέθηκε σήμερα είναι καινούρια. Όπω είπε πολύ σωστά και ο εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου, θα πρέπει να εξετάσουμε τη σχεση κοστους κόστου-οφέλου ε, και να βρούμε μια κατάλληλη ισορροπία για να υπάρχει και καλής ποιότητας πραγματογνωμοσύνη ε, και ανεξαρτησία στο ενύψιστο δυνατό βαθμό και είναι λοιπόν μια πρόταση που θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά μαζί με την ΕΦΣΑ. Και να επιβεβαιώσω, όπω είπε και ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή σήμερα το πρωί, ότι σε ό,τι αφορά τη σύσταση για την σύσταση ε, κοινού ε, πλαισίου για την εξαρτησία των οργανισμών. Είναι μια σύσταση που έγινε και από την ε, διοργανική ομάδα για τους οργανισμούς που συμπεριλήφθηκε στον οδικό χάρτη της Επιτροπής τις ε, ενέργειες 33 και 35. Είναι λοιπόν ένα εγχείρημα που έχει ξεκινήσει η Γενική Γραμματεία και αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές θα υιοθετηθούν μέχρι τα τέλη του 2013. Και είναι ένα εγχείρημα που θα ε, λάβει χώρα και σε συνεργασία με τους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Φτάνουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα τη ημερησία διάταξη που είναι η οδηγία για το μέλη και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια την κυρία Γκέρλινγκ. Παρακαλώ. Thank you. This one's working. Um, I'm just going to uh, run through uh, briefly, very... Ευχαριστώ πολύ. Θα διατρέξω εν συντομία την έκθεσή μου και τη θέση μου σε αυτήν. Είναι μια σχετικά απλή έκθεση. Η Επιτροπή είχε δύο λόγους για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Πρώτος λόγος είναι η διευκρίνηση του νομικού καθεστώτος ε, της γύρισης και του μελιού μετά την ε, απόφαση του δικαστηρίου που λέει ότι ε, η γύρη είναι συστατικό του μελιού και δεύτερον για την ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Εθνικής Λισαβόνας για τις κατεξουσιοδότηση πράξη. Για το πρώτο, λοιπόν, η απόφαση του δικαστηρίου του Σεπτεμβρίου του 2011 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέλι που ε, συμπεριλαμβάνει ε, γενικά τα τροποποιημένη γύρι θα πρέπει να θεωρείται ω ε, τρόφιμο που βάσει τα τρόφιμα που υπάγονται στα γενετικά τροποποιημένα. Και έτσι ε, θεωρείται ότι είναι συστατικό η γύρι του μελιού. Η πρόταση της Επιτροπής ε, αμφισβητεί αυτή την ε, θέση. Λέει ότι είναι ε, στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, όχι συστατικό. Και αναφέρεται και στον ορισμό του μελιού ότι δεν συμπεριλαμβάνει συστατικά. Αυτό είναι ο βασικός όρισμος που υπάρχει, ότι η γύρι είναι στοιχείο της σύνθεσης του μελιού και όχι συστατικό. Όλο το επιχείρημα βασίζεται σε αυτό λοιπόν. Για αυτούς τους λόγους και έχοντας εξετάσει όλα τα στοιχεία και έχοντας συζητήσει με εκπροσώπους αδιαφόρων ε, ομάδων ενδιαφέροντος, εγώ θεωρώ ότι συνάδει με τον κόντεξ και σε αυτό συμφωνούν και οι καταναλωτές, ότι δηλαδή το mail είναι ένα και μοναδικό προϊόν. Δεν ε, είναι ένα αμάλγαμα διαφορετικών ε, συστατικών. Γι' αυτό και με τα χαράς ε, δέχθηκα αυτό το τμήμα της πρότασης της Επιτροπής με ίσονο σημασία τροπολογίες, όπως θα δείτε και από την έκθεσή μου. Επομένω, δεν θεώρησα ότι θα έπρεπε να τροποποιηθούν πολλά, εφόσον συνάδουν, όλα αυτά και με τα όσα κάναμε εμείς πρόσφατα στην Επιτροπή μας για την πληροφόρηση των καταναλωτών. Τώρα, σε ό,τι φορά όμως ε, την ευθυγράμμιση υπάρχουν κάποια σημεία πήρα την θέση παρόμοια με αυτήν που υπήρξαν στις οδηγίες ε, ε, περί του προγεύματος. Εκεί πέρα λοιπόν ε, ε, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή μέσω καταξιδότηση πράξεων ε, για τα ονόματα των προϊόντων, κριτήρια σύνθεση, τα στοιχεία που διασφαλίζουν ότι αυτό που αγοράζουμε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επισήμανση μελιού, ότι είναι πράγματι μέλη και διασφαλίζεται έτσι και η ακαιρεότητά του θεωρώ ότι είναι θεμελιώδη στοιχεία της ε, ε, οδηγίας γιατί καθορίζουν τι ακριβώς μπορεί να τεθεί σε εμπορία και να αποκληθεί μέλη. Σύμφωνα με τη συνθήκη, ο νομοθέτης μπορεί να δώσει τέτοιες ε, εξουσίες στην Επιτροπή μόνο για τα μη ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας. Γι' αυτό στις τροπολογίες μου εγώ έχω διαγράψει το πεδίο εφαρμογής σε ό,τι αφορά τα παραρτήματα, αυτά έβγαλα. Λοιπόν, οποιαδήποτε τροποποίηση των παραρτημάτων θα πρέπει να περνάει από την συνήθη νομοθετική διαδικασία. Για να θίξουμε ελαφρώς αυτό το, ζήτημα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, ε, η πρόταση της Επιτροπής προτείνει να δεχθούμε την πρόταση του, μελιού... του δικαστηρίου για το μέλι, μέλι, όπως συμβαίνει και σε άλλα τρόφιμα. Εγώ συμφωνώ. Και πάλι θεωρώ ότι δεν χρειάζονται άλλες ε, τροπολογίες. Ε, με συζητήσεις ε, με σχιώδη, που βέβαια έγιναν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατάλαβα ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες και προβληματισμοί από αυτού. Κατά τη διάρκεια τη σημερινή συνεδρία σα ελπίζω να ε, βρούμε κοινό έδαφος. Äh, e Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χίπνερ εκπροσωπείται το ΕΛΚΑ. Για τους σοσιαλδημοκράτες, Λίντα Μακέβεν. Yes, I'm my colleague... Um... Ναι. Η κυρία Ταβάζη, εσύ συνάδελφος, μου ζήτησε να διαβάσω το κείμενο της στην Επιτροπή σας. Σχετικά με την ε, ιδέα της μεταστατικής τύπου, Λέει λοιπόν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Βαβαρία έναντι και Παπλόκ, Ένωση Μελισσουργών, χύνει φως στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί γενετικά τροποποιημένων. Σε αυτή την περίπτωση η έλλειψη αναγκαστικών μέτρων οδήγησαν στην επιμόλυνση του μελιού με γενετικά τροποποιημένη γύρι, κάτι που δεν μπορεί να δοθεί σε ανθρώπινη κατανάλωση. Σοβαρό ζήτημα που απαιτεί εξέταση και ρυθμιστικές απαντήσεις. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει είναι μόνο για τεχνική λύση. Αντίθετα στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και λέει ότι οι γύροι θα πρέπει να τι, φυσικό συστατικό του μελιού και όχι ε, υλικό στη σύνθεση του μελιού. Constituents στα αγγλικά και όχι ingredient. Αν συμβαίνει αυτό, τότε ξεπερνούμε τον κανονισμό περί γενετικά τροποποιημένων, καθώ η συγκέντρωση γύρι πρέπει να πάτε κάτω από το 0,5% στο μελιό. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα φτάνουμε το κατόφλι του 0,9% για κάτω πεπιμένο, οπότε πάνω από αυτό θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του καταναλωτή στην ετικέτα. Αποτέλεσμα αυτού, η πρόταση θα πρέπει να υιοθετηθεί με την... αν υιοθετηθεί στην παρούσα μορφή θα οδηγήσουμε σε παραπλάνηση του καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο δεν αντιμετωπίσετε το σοβαρό και υφιστάμενο πρόβλημα που είναι ότι δεν έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία εν προκειμένου. Γι' αυτό ε, η ομάδα σολιστών ζήτησαν μελέτη δικτύπου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αρμόδια του υπηρεσία και να αναβληθεί η ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών σε αυτή την έκθεση ως συνέπεια αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Ράιμας είναι σκιώδη συγγήτρια των Φιλελεύθερων. Έχει τώρα το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι διάβασα προσεκτικά την πρόταση της κυρίας Κέρλινγκ ε, και νομίζω ότι πρέπει να την υποστηρίξουμε. Η γύρι είναι ακριβώς στοιχείο και όχι συστατικό του μελιού. Από την απόφαση του δικαστηρίου προκύπτει ο τρόπος χειρισμού του θέματος. Υπάρχει νομική ανασφάλεια διότι η ε, παραγωγή μελιού δεν ε, ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και δεν ε, υπάρχει μια αξιόπιστη διαδικασία όσον αφορά την ε, γενετικά τροποποιημένη γύρη και αυτό σημαίνει ότι η απόφαση του ε, δικαστηρίου δεν είναι εφαρμόσιμη. Εάν δηλαδή θα πρέπει να αποδειχθούν όλα αυτά θα είναι τεράστιο το κόστος και αυτό δεν είναι στόχος κανενός. Ε, εάν θεωρήσουμε ότι η γύροι ούτως ή άλλως ε, ε, περιλαμβάνεται στο μέλι σε ποσοστό μικρότερο του 1%, Νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη ζημιά και για τους μελισσοκόμους αν πρέπει να το αναγράφουν αυτό. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η προσαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας Έχουμε τώρα πια την συνηθισμένη ε, διαμάχη με την Κομισιόν ε, σχετικά με τις αρμοδιότητες. Ο καθένας ερμηνεύει με τον τρόπο του τη συνθήκη της Λισαβόνας και θα ήθελα ε, να συμφωνήσω και με την ερμηνεία της συνθήκης που περιλαμβάνεται εδώ. Όσον αφορά την μελέτη αντικτύπου, και αναβολή της απόφασης. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε, διότι εάν ε, θέλουμε να κάνουμε μια ε, μακροπρόθεσμη ε, έρευνα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημίες για τους μελισσοκόμους, διότι κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να περιλαμβάνεται στην επισήμανση αυτή τη στιγμή. Εάν πρόκειται να κάνουμε μελέτη αντικτύπου, θα πρέπει να Ε, σκεφτούμε ότι οι επιτόπου εμπειρογνώμονες ε, έχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Θέλουμε να ε, φροντίσουμε να μην επιφέρουμε επιπλέον δαπάνες με τα αιτήματά μας για επιπλέον έρευνες. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με την κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ράιμερ. Ο Μπάρστας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν νομοθετούμε βεβαίως ε, δεν ε, νομοθετούμε από ε, τον υψηλό μας πύργο. Από την συνάντηση των σκιωδών εισηγητών που έλαβε χώρα στη, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας το Δεκέμβριο, τότε μόνο συναντηθήκαμε με τους σκιώδεις, υπήρχε ακόμα μια βεβαιότητα για τη θέση των, των ενδιαφερομένων μερών από αυτής της πρότασης. Και τότε είχα έρθει σε επαφή με εκπροσώπους από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Και τότε στην ε, συνάντηση των σχεδόν είχα ζητήσει από την εισηγήτρια μήπως ε, την είχα ρωτήσει μήπω θα ήταν καλό και σκόπιμο να υπάρξει αξιολόγηση αντικτύπου. Γιατί τουλάχιστον από αυτέ τι δύο μεγάλε χώρε υπήρχε σημαντικό προβληματισμό. Εν τω μεταξύ υπάρχει και κοινή θέση 19 οργανισμών από 11 χώρε. Δεν είναι και ασήμαντο αυτό και μικρότερε και μεγαλύτερε χώρε. Όμω είναι ε, σημαντική, ε, σημαντικός ο κατάλογος από Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Μάλτα, Ουγγαρία, Κύπρος, ε, Ισπανία, μεταξύ άλλων. Έτσι. Και όλες αυτές οι οργανώσεις είναι κατά της ε, ε πρότασης, γιατί θεωρούν ότι ο, αντίκτυπος ε, της πρώτης επιτροπής θα είναι πολύ αρνητικός στις ε, δραστηριότητές τους. Είναι μια περίεργη κατάσταση, συνάδελφοι, γιατί πώς ξεκίνησαν τα πράγματα. Ακριβώς επειδή ένας ε, αριθμό φορέων από τη Γερμανία ε, ανησυχούσε για αυτήν την κατάσταση, ξεκίνησε μια δικαστική υπόθεση που έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλοι ε, χάρηκαν με την απόφαση γιατί υπήρξε βεβαιότητα και τώρα υπάρχει μια νέα πρόταση της Επιτροπής που δημιουργεί εκ νέου ανασφάλεια. Και έτσι συμφωνώ με το ερώτημα των σοσιαλιστών αλλά και με τον κύριο Πετριλέ ε, για το αίτημα για αξιολόγηση δικτύπου. Εφόσον τόσε οργανώσει οργανώσεις το έχουν ζητήσει, νομίζω ότι είναι δόκιμο. Και από τότε, από την τελευταία συνάντηση, είπε η συγκήτρια ότι ε, επικοινωνούσαμε μέσω email, αλλά αυτό ήταν επικοδοματικό και σας ευχαριστώ που πάντα απαντούσατε τόσο γρήγορα και με καλή διάθεση. Εάν ε, πρέπει να γίνει εξολόγηση δικτύπου, τότε θα πρέπει να απαντηθούν κάποια ερωτήματα. Ε, αν το μέλι θεωρηθεί φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι αυτό θα σημαίνει και για, την, ε, για τις υποχρεώσεις σήμανσης ε, υπό την νομοθεσία για τα τρόφιμα και για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δεύτερον, ποιες επιπτώσεις έχει αυτό ε, στην νομοθεσία ε, στα κράτη-μέλη για την αποζημίωση αν, υπάρχουν, ε, αν υπάρχει γενετικά τροποποιημένη γύρι μέσα στα μέλη. Δεύτερον, ποιος θα είναι ο, αντίκ, τρίτον, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος ε, στις, ε, στους ε, μελισσουργούς και στις οικονομικές δραστηριότητες και η ενδεχόμενη απώλεια εμπιστοσύνης ε, από τους πολίτες σε ένα τέτοιο καταπληκτικό φυσικό προϊόν όπως είναι το μέλι. Τέταρτο ερώτημα. Ποιος θα είναι αρνητικός αντίκτυπος στη γεωργία και στα οικοσυστήματα. Και τέλο, υπάρχει και το ερώτημα ποια, ποιες θα είναι οι επιπτώσει αυτή τη πρόταση στη διαφάνεια. Επιπλέον, ε, ρητό ερώτημα προς την Επιτροπή. Βλέπω ότι είναι εδώ και η κυρία Μπουτλέ. Πολύ φοβάμαι ότι ε, παραβλέπουμε μια ενδεχόμενη λύση. Υπάρχει μια εναλλακτική λύση κατά τη γνώμη μου. Αν εξετάσουμε την νομοθεσία σήμανσης ε, τροφίμων, όπου υπάρχει δυνατότητα κατάρτισης καταλόγου ε, καταλόγων ε, προϊόντων τροφίμων τα οποία θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο συστατικών το τυρί, για παράδειγμα, βρίσκεται ε, σε αυτά τα προϊόντα, σε ένα τέτοιο κατάλογο. Και εκεί πέρα δεν ε, εφαρμόζονται αυτέ οι διατάξει. Αν βάλουμε το μέλι σε αυτόν τον κατάλογο, τότε ο αρνητικό αντίκτυπο όλη τη πρόταση για του μελισσουργού ε, αποφεύγεται. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά, πολλοί άριθμα ερωτήματα για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε. Συμφωνώ ακριβώς όπως πολύ σωστά έθεσε αυτό το ερώτημα ο κύριος Σταμπάτζη στο κείμενο που ε, διάβασε η συνάδελφος προηγουμένως και οι πράσινοι καθώς και οι σοσιαλιστές και ε, άλλες ομάδες ε, ρωτούν μήπως θα έπρεπε το Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει μια τέτοια αξιολόγηση δικτύπου. Νομίζω ότι συζητήθηκε και σήμερα το πρωί στην συνάντηση των συντονιστών ότι υπάρχει έλλειψη χρόνου, ωστόσο θα ήθελα ε, να καλύψω τους συναδέλφους να αντιδράσουν θετικά. Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το δικαστήριο ήθελε να εγγυηθεί πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή. Αυτό πώς το θέραπε πέρας με την ετικετοθεσία στα τρόφιμα. Αυτό που δεν προβλέψαμε είναι αυτό το, πρόβλημα. Τι είναι φυσικό στοιχείο ε, ενός ε, τροφίμου και που άρα δεν μπορεί να διαχωριστεί, δεν είναι υλικό πρόσθετο. Το μέλι λοιπόν δεν αποτελείται από διάφορα υλικά, αλλά από φυσικά συστατικά που δεν μπορούν να διαχωριστούν από το προϊόν που είναι το μέλι. Και εδώ ήταν το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Άρα, τώρα το δικαστήριο αποφασίζει ότι το μέλι μπορεί όμως να υποδιαιρεθεί σε επιμέρους υπομονάδες, υποσυστατικά. Ε, δεν είναι όμως σωστό αυτό. Θα πρέπει να το δούμε το θέμα από ένα άλλο πρίσμα. Γιατί θα καταλήξουμε σε κάτι τελείως παράλογο. Το εν λόγω προϊόν, αν είναι ε, το όλον και δεν μπορεί να, να, να, να υποδιαιρεθεί, τότε εμείς έχουμε δίκιο και αυτός μιλάμε για ένα φυσικό συστατικό. Αν κάνουμε τέτοια υποδιέρεση θα κάνουμε κάτι τεχνητό και κάτι λανθασμένο. Γι' αυτό υποστηρίζω την εισηγήτρια. Θέλουμε να βγάλουμε τελείως εκτός αυτό το κλάδο της μελισσουργίας. Ε, θέλουμε πλήρη ενημέρωση στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους γενικά τροπημένους, αλλά να μην μπαίνουμε σε κάτι παράλογο. Ευχαριστώ, Εκπλήσουμε από τα όσα υπόθηκαν σήμερα ότι ε, η απόφαση του Δικαστηρίου ε, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι παράλογη. Ε, είχα δύο πράγματα να πω. Πρώτα απ' όλα δεν θεωρώ ότι ο στόχος είναι να στραφούμε εναντίον του, της απόφασης του δικαστηρίου, απλώς να αντλήσουμε συμπεράσματα από αυτήν. Δεύτερη παρατήρηση, συμφωνώ πολύ με τα όσα είπε ο και με τα όσα είπε συναδελφό μας. Ε, νομίζω ότι αν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους γεωργούς και να τηρήσουμε και τις αποφάσεις του δικαστηρίου πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητη μια αξιολόγηση αντικτύπου γιατί δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ε, τα στοιχεία στην οποία βασίστηκε, ε, στην οποία βασίστηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι δεν μπορούμε να στραφούμε κατά της. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ε, πρόσεξα τον συνάδελφο, του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, και εγώ συμφωνώ με όσους ε, αναρωτιόνται αν αξίζει τον κόπο ε, να διαφωνήσουμε με την απόφαση ε, του δικαστηρίου και να θεωρήσουμε ότι το μέλι είναι στοιχείο και όχι συστατικό του μελιού. Το θέμα από την πλευρά ε, του καταναλωτή είναι αν το μέλι περιέχει πάνω από 0,9% γενετικά τροποποιημένης γύρης. Και πιστεύω ότι η απόφαση του δικαστηρίου και η προσέγγιση του δικαστηρίου είναι καλή. Ε, και όσον αφορά την επισήμανση. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε όμως ε, τι θεωρούν οι Ευρωπαίοι μελισσοκόμοι, οι οποίοι συμφωνούν απόλυτα με την απόφαση του δικαστηρίου. που θεωρεί ότι η γύρι δεν είναι συστατικό του μελιού. Νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την ε, εισαγωγή μελιού από τρίτες χώρες, διότι αν κοιτάξουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή, τότε διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος ε, του μελιού ε, που κυκλοφορεί προέρχεται από χώρες όπου ε, δεν ε, υπάρχει μολυσμένο, χιον, ε, μέλι, μολυσμένο μέλι με ε, ποσοστό γενετικά τροπημένων οργανισμών άνω το 0,9% προέρχεται από τις ε, χώρες της Λατινικής Αμερικής για παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι δεν νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τις ε, ξένες ε, μάρκες. Ε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε μελέτη επιπτώσεων και κατόπιν να διαπιστώσουμε αν η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να υποστηριχθεί από τους εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ. Ε, ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Θα ήθελα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, παρακαλώ. Να ζητήσω συγγνώμη κιόλα ε, που δεν είχαμε θέσει για να καθίσετε. Ε, αυτό οφείλεται στο ότι δεν είμαστε στην ε, δικιά μα αίθουσα, στην αίθουσα που χρησιμοποιούμε συνήθως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κανένα πρόβλημα δεν υπήρξε που σταθήκαμε και όρθιοι για μερικά λεπτά. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκέρλινγκ για την έκθεσή της. Την ευχαριστώ θερμά γιατί η έκθεση κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης ε, Καταναλωτών. Ε, και αν με επιτρέπετε και η Γενική Διεύθυνση, ο Γενικός Διευθυντής της ε, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας θα μπορεί να απαντήσει για το τμήμα που αφορά τις συνθήκες της Λισαβόνας. Σας επιστρέψω τώρα στο μέλη και στη γύρι. Συμμεριζόμαστε την θέση της κυρίας Λεπάζ ότι δηλαδή δεν μπορούμε να επικρίνουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεχόμαστε ε, τις αποφάσεις ε, του δικαστηρίου χωρίς κανένα πρόβλημα. Το δικαστήριο σε αυτή την απόφαση απέστειλε μια απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα του γερμανικού δικαστηρίου που του έθεσε αυτό το ζήτημα. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ερμήνευσε ε, βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Υφιστάμενης υπογραμμίζω. Και πράγματι η υφιστάμενη νομοθεσία, η οδηγία για το μέλη, δεν ήταν σαφής σε αυτό το σημείο. Και υπήρχε θέμα προς ερμηνεία και το δικαστήριο θεώρησε ότι η γύρι αποτελεί συστατικό ingredient. Όμως, ε, όπως όλοι οι επιστήμονες αναγνωρίζουν, η γύρι δεν είναι στατικό, δεν προστίθεται από τον μελισσοκόμο ε, κατά την ε, επεξεργασία του μελιού. Η γύρι είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης. Γι' αυτό βρίσκεται στις αρμοδιότητες και στις εξουσίες του νομοθέτη να τροποποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία για να διευκρινίσει κάτι που δεν ήταν σαφές στην προηγούμενη νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε να παρακάμψουμε την απόφαση του δικαστηρίου καθόλου. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό την αποδεχόμαστε. Το δικαστήριο λέει ότι ε, οποιαδήποτε νομοθεσία για τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ε, εφαρμόζεται και για την γύρι σε ό,τι αφορά την ετικετοθεσία. Την εφαρμόζουμε, όπως και στο παρελθόν είχε εφαρμοστεί, επειδή λέγαμε ότι είναι, η γύρι είναι προϊόν ζωικής προέλευσης και δεν μας αφορούσε εκείνη την περίοδο. Το υιοθετούμε λοιπόν και προτείνουμε εδώ να διευκρινίσουμε ότι η γύρι είναι φυσικό στοιχείο και όχι συστατικό. Δεν παρακάμπτουμε έτσι λοιπόν την απόφαση του δικαστηρίου, απλώς διευκρινίζουμε με μια νέα πρόταση ότι ο νομοθέτης, δηλαδή εσείς και το Συμβούλιο, ε, είναι, έχουν δικαίωμα να το πράξουν έτσι κι αλλιώς. Εδώ σημαντικό είναι ότι έρεται η αβεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχει μια αβεβαιότητα. Γιατί ιδίω η ε, οι γύροι ε, της Μονσάτο 810 του Αραβοσίτου μέχρι τώρα δεν ε, είχε λάβει αδειοδότηση. Έχουμε ζητήσει από την ΕΦΣΑ να κάνει μια γρήγορη αξιολόγηση για να δει αν αυτή η γύρι παρουσιάζει κινδύνους, έχει κινδύνους για το περιβάλλον, για τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ε, μελισσών ε, και ούτω καθεξής. Η ΕΦΣΑ απάντησε αρνητικά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και ζητήσαμε από τη Μονσάντο να υποβάλει αίτημα για να αξιολογηθεί από την ΕΦΣΑ αυτή η γύρη και να αδειοδοτηθεί, αδειοδοτηθεί επισήμως. Και έτσι έρεται η αβεβαιότητα. Αυτό συνέβη λοιπόν. Βεβαίως το πρόβλημα της, ε, του, του εισαγόμενου μελιού υφίσταται και αυτό γιατί ε, υπάρχουν μη γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί που ε, δεν αντιδοτούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αντιδοτούνται σε τρίτες χώρες και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Για τον Καναδά, για την Αργεντινή που εξάγουν μέλι γιατί εμείς εισάγουμε 50% του μελιού που καταναλώνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παράγουμε το 50% και εισάγουμε το υπόλοιπο 50%. Οι εισαγωγέ ε, αφορούν κυρίω ε, ε, τη, τη βιομηχανία, δηλαδή τη ζαχαρο, ζαχαροπλαστική που χρησιμοποιεί μέλι. Αλλά και από τι βιομηχανίε που το επεξεργάζονται για να το τρώμε εμεί στο, στο πρωινό μα. Αλλά και από ε, τον τομέα των ε, καλλιτικών. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η πρόταση διευκρινίζει την κατάσταση και το καθεστώς ε, της γύρης που αποτελεί φυσικό στοιχείο και μετά ο κανόνας προφανώς της ετικετοθεσίας για τα γενικά τροποποιημένα εφαρμόζεται με το κατόφλι του 0,9% όπως γνωρίζετε. Δηλαδή το μέλι θα πρέπει ε, να έχει ετικέτα. Αν έχει πάνω από 0,9% γύρις, ε, γενετικά τροποποιημένης γύρις. Βεβαίω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε ότι όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει λιγότερο από 0,9% γύρι ε, στο μέλι. Από το 0,1 μέχρι 0,4% maximum. Επομένως, δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι ε, είναι μάλλον απίθανο να υπάρχει ετικέτα όταν υπάρχει γύρι ε, γενετικά τροποποιημένη, γιατί δεν ξεπερνά η γύρι αυτή την ποσότητα. Όμως ο κανόνας εφαρμόζεται, ενώ προηγουμένως ε, λανθασμένα, και το αναγνωρίζουμε εφόσον μας το είπε το δικαστήριο, ότι δεν εφαρμοζόταν. Αυτή είναι μια παρατήρηση που θέλω να κάνω. Τώρα, μια απάντηση προ τον κύριο Στάση για την εναλλακτική του που προτείνει. Μα το να χρησιμοποιήσουμε τον κατάλογο των αισθητικών που είναι απαγορευμένα και δεν πρέπει να υπάρχουν σε ένα τρόφιμο. Ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό, αυτή τη διάταξη της νομοθεσίας για την ετικετοθεσία των τροφίμων. Όμως αυτό σημαίνει ότι η γύρι ε, γίνεται συστατικό μετά. Όμως ολόκληρη αυτή την προσπάθεια την κάνουμε για να πούμε ότι δεν είναι συστατικό γύρι, είναι φυσικό στοιχείο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διάταξη, όμως αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε, όπως είπε το δικαστήριο, ότι η γύρι είναι συστατικό. Και δεν συμφωνούμε με αυτό. Οι ίδιοι επαγγελματίες γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για στατικό αλλά για φυσικό στοιχείο. Δυστυχώ, λοιπόν η πρόταση του κυρίου Στάς δεν μπορεί να ε, αξιοποιηθεί ως εναλλακτική λύση. Δεν, να πούμε δηλαδή ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γύρι γενετικά τροποποιημένη προέλευση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η μοναδική νομοθεσία που εφαρμόζεται που, για, για τη γύρι, τη γενικά τροπημένη γύρι στο μέλι είναι με αυτό το κατόφλι του 0,9% που κατά πάσα πιθανότητα, όπω ξέρετε, δεν θα φτάσει, ε, δεν θα, η υπερεκτικότητα του μελιού σε γύρι δεν φτάνει το 0,9%. Ε, να επιτρέψουμε τη συνάδελφο, το, το συνάδελφο από την άλλη Γενική Διεύθυνση να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. σε ό,τι αφορά την πρόταση τη Επιτροπή για την ευθυγράμμιση με του νέους κανόνες Επιτροπολογία ε, για τις συνθήκε τη Λισαβόνα, ε, να πούμε μόνο ότι, όπω είπε και η κυρία Γκέρλινγκ, αλλά και άλλοι ευρωβουλευτέ, είναι ένα ζήτημα σημαντικό που δεν έχουμε πάντα την ίδια προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων, δηλαδή ε, τον ε, προσδιορισμό ε, και την ταξινόμηση των εξουσιών της Επιτροπής, δηλαδή ανάμεσα σε καταξιδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Πρέπει να δούμε, δηλαδή, με ποια προσέγγιση ε, εκπονήθηκε αυτή η πρόταση. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι οι εξουσίες που συμπεριλαμβάνονται, που προτείνονται δηλαδή εδώ στο κείμενο, είναι υφιστάμενες εξουσίες ε, βάσει της ε, υπάρχουσας οδηγίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 σε τη τη μέθοδο ανάλυσης και στο άρθρο 6 για την δυνατότητα της Επιτροπής να προσαρμόσει ή να συμπληρώσει τα περαρτήματα 1 και 2 της οδηγίας για το μέλη. Και πρέπει να προσδιορίσουμε ότι οι εξουσίες που προτείνει η Επιτροπή στο νομοθέτη να τις εκχωρηθούν, μπορούν να περιοριστούν. Εφόσον σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόθεση της Επιτροπής να τροποποιήσει ε, ουσιώδεις επιτυχές ε, των παραρτημάτων αυτών. Απλώς θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε, να συμπληρώσουμε ε, στοιχεία τεχνικής φύσεως που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα δύο παρατήματα και αφορούν τις, τις περιγραφές, ε, την αναπαράσταση και την ονομασία ε, αυτών των προϊόντων μελιού. Επομένω, Πρόεδρε, θεωρούμε ότι οι εξουσίες ε, που προτείνουμε να μας εκχωρηθούν για να τροποποιήσουμε την οδηγία ε, αφορούν ε, την, αποφασιστη... την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα της νομοθετικής διαδικασίας και για τα απολύτως τεχνικά ζητήματα και για την προσαρμογή μας στο πλαίσιο του ε, Διεθνούς Ομοθετικού Πλαισίου και του Κόντεξ Ελεμαντάριου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τέθηκε μια ερώτηση σχετικά με τη ε, μελέτη αντικτύπου από τον συνάδελφο Μπάρτστας. Σήμερα το πρωί στους ε, συντονιστές ε, είπαμε ότι θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό και στην Επιτροπή για να υπάρχει διαφάνεια μελέτη αντικτύπου από την Κομισόν θα διαρκέσει κανένα χρόνο ε, μέχρι να τη δούμε, ενώ η δική μας ε, μπορεί να γίνει πιο γρήγορα, μέσα σε τέσσερις μήνες ε, είναι το πιθανότερο. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. θα πρέπει να το, να το συζητήσουμε. Βέβαια, τίποτα δεν είναι δωρεάν, αυτά στοιχίζουν, αλλά η δημοκρατία στοιχίζει. Η συγγήτρια, κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω αναλυτικά σε όλα, αλλά να συνοψίσω ποια πιστεύω εγώ ότι είναι τα σημαντικά θέματα. Το όλο θέμα έχει να κάνει με τον ορισμό, όπως σας είπα. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και να μην μπερδευτούμε με όλα τα άλλα θέματα, τα οποία μπορεί να είναι πραγματικές ανησυχίες. Πράγματι είναι πραγματικές ανησυχίες, αλλά δεν σχετίζονται με την απόφαση αυτή. Μία μελέτη αντικτύπου θα έχει να κάνει με την αλλαγή των, κανόνα. Αυτή τη στιγμή, των κανόνων. Αυτή τη στιγμή έχουμε την οδηγία για το μέλη, έχει δημιουργηθεί νομική αβεβαιότητα λόγω μιας απόφασης ε, του δικαστηρίου, αλλά η τροποποίησή μας θα μας φέρει στο status quo αυτή τη στιγμή. Δεν θα γίνει κάποια σημαντική αλλαγή. Αυτό ήταν όλο το θέμα όσον αφορά τον αντίκτυπο. Ναι, θα υπάρχει αντίκτυπος για τους μελισσοκόμους. Αλλά, εκεί είναι δύσκολο να το εξηγήσω αυτό, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει αντίκτυπο, δεν θα αλλάξει τίποτα για κανέναν που παράγει ή πουλάει το μέλι. Γι' αυτό ακριβώ δεν έγινε μελέτη αντικτύπου και γι' αυτό η αρχική μου αντίδραση ήταν ότι δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητη μια μελέτη αντικτύπου. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στον κύριο Τοπαίδη μέσω της Λίντα ε, όταν μίλησε για παραπλανητική επισήμανση. Δεν καταλαβαίνω πώς συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί ουσιαστικά τίποτα δεν αλλάζει. Αν ένας ε, παραγωγός, ε, θέλει να γράψει ότι το μέλι του είναι απειλαγμένο από γενετικά τροπημένους οργανισμούς, μπορεί να το κάνει αυτό, τίποτα δεν αλλάζει. Το θέμα εδώ είναι τα όρια για την επισήμανση, αλλά αυτό δεν ε, έχει να κάνει με την, ε, ε, με την οδηγία του μελιού. Μπορεί να με βρίσκει σύμφωνη το θέμα αυτό, αλλά δεν έχει τη θέση του σε αυτή την οδηγία. Επίσης, αρκετοί ομιλητές είπαν ότι οι μελισσοκόμοι δεν συμφωνούμε με την πρόταση της Κομισιόν. Ενώ γνωρίζω ότι ο κύριος Στές και άλλοι μπορούν ε, Μπορεί να έχουν λίστες με, κατα... που διαφωνούν, ε, αλλά εγώ μπορώ να σας δώσω παραδείγματα ενώσεων ε, μελισσοκόμων ε, που είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με την πρότασή της Κομισιόν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να παίξουμε το παιχνίδι των αριθμών, ποιο είναι υπέρ και ποιο είναι κατά, διότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Υπάρχουν ανάμεικτες ε, απόψεις και πολλές ενώσεις μελισσοκόμων μου είπαν ότι ειλικρινά δεν βλέπουμε πού υπάρχει πρόβλημα. ενώ άλλοι μου έκαναν ε, πολύ σημαντικά παράπονα, αλλά ε, δεν ε, έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη πρόταση. Όσον αφορά την εναλλακτική πρόταση του κυρίου Στάς, μπορώ να πω ότι την εξέτασα προσεκτικά πριν γράψω την έκθεσή μου, πήρα και νομικές συμβουλές και κατέληξα στο ίδιο ε, συμπέρασμα ότι δεν θα ήταν ε, βιώσιμη η μέθοδος αυτή, θα μπορούσε ε, να προβληθεί νομικά και θα οδηγούσε στη συνέχιση της νομικής ανασφάλειας. Ε, ζητώ συγγνώμη που ξέχασα να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές ε, για την βοήθειά τους, αλλά το συμπέρασμα μου είναι ότι δεν είναι απαραίτητη μια μελέτη αντικτύπου. Ωστόσο, ε, σημειώνω τις ανησυχίες. Έχω συνομιλήσει με μεριστοκόμους σε όλη την Ευρώπη και καταλαβαίνω κάποιες από τις ανησυχίες τους. Όμως, θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι ο λόγος που η Κομισιόν χρειάζεται 12 μήνες ε, είναι ότι μεγάλο μέρος ε, του διαστήματος αυτού είναι διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους. Αν είναι να κάνουμε διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, νομίζω θα πρέπει να γίνει σωστά ε, και αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και συνεργασία των ενδιαφερομένων και διαβούλευση. Εάν επιλέξουμε τη μέθοδο του Κοινοβουλίου, αυτό δεν θα γίνει. Λοιπόν, θέλουμε είτε πλήρη διαβούλευση ή τίποτα. Αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Θα παρακαλούσα όλους να το σκεφτούν και να σκεφτούν και τι συνέπειε. Μιλήσατε για ε, νομική ανασφάλεια με μια καθυστέρηση των δεκαμήνου και νομίζω ότι ε, αυτό θα ε, βλάψει αρκετούς οι μελισσοκόμοι. Λένε ότι σα παρακαλώ μην το κάνετε αυτό, θέλουμε να κλείσει το θέμα τώρα. αν κάποιος θέλει να μιλήσει μαζί μου πριν την επόμενη συνεδρία των συντονιστών για το θέμα της μελέτης αντικτύπου, πολύ ευχαρίστως μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκέρλινγκ. Έχουμε την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, ε, ε, την έχουμε μεταφέρει στις 21 Φεβρουαρίου 12 η ώρα. Και στους συντονιστές ε, θα, μιλήσουμε, θα συζητήσουμε το θέμα της ε, μελέτης αντικτύπου. Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και προχωράμε τώρα στο σημείο 28 της ημερησίας διάταξης. Έχουμε και εδώ προφορική ερώτηση του Chris Davis. Θα ήθελα λοιπόν να του δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Chris Davis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να δώσουμε πρώτο το λόγο στην Κομισιόν και μετά να κάνω συμπληρωματικές ερωτήσεις. Ε, η Κομισιόν έχει το λόγο, παρακαλώ. Oui, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόβλημα των νέων νοικοτενοειδών είναι σοβαρό και σημαντικό. Για την υγεία των μελισσών, επιτρέψτε μου να το πω για να συνδέσω και τα δύο ζητήματα με το προηγούμενο. Είναι πολύ πιο σοβαρό λοιπόν από τη γύρι ε, της Μονσάντο. Ε, το πρόβλημα των νέων νοικοτενοειδών δεν είναι πρόσφατο οι ίδιοι οι μελισσοκόμοι είχαν ιδιαίτερε επιφυλάξει για, το, για αυτά τα προϊόντα για πάνω από μια δεκαετία τώρα. Εμείς ειδοποιήσαμε ε, την ΕΦΣΑ πριν από πέντε χρόνια περίπου για αυτό το πρόβλημα. Το 2010 υιοθετήσαμε οδηγία της Επιτροπής για την ενίσχυση των μέτρων που υιοθετούν, ε, ε, υιοθετεί η βιομηχανία ε, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των νέων και βεβαίως το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί με την, ή μάλλον έχει επιταχυνθεί η μαλλον εχει επιταχυνθει τη διαδικασια με τις δύο μελέτες, μία γαλλική και μία βρετανική και μία τρίτη γερμανική την τελευταία χρονιά, το Μάρτιο του 2012. Και σε αυτές τις ε, μελέτες φάνηκε ότι οι πολύ μικρές δόσεις των νοικοτινοειδών απατώντας τα λουλούδια, στα άνθη, ε, στα φυτά των οποίων οι σπόροι ε, είχαν τύχη επεξεργασία με νέο ε, τον οποίο τον νέκταρ παίρνουν οι μέλισσες για να παράξουν το μέλι. Έχουν όμως μια μη θανατηφόρα βέβαια τοξικότητα δεν πέθανε δηλαδή κατευθείαν οι μέλισσες, Όμω ε, ε, αποπροσανατολίζονται, δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Κυψέλη. Όπω συμβαίνει Δηλαδή δεν ήταν θανατηφόρε οι δόσει όπω συμβαίνει με άλλα ζυζανιοκτώνα που απαγορεύεται ε, να ε, χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο τη άνθηση. Αυτό είναι σημαντικό γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 80% των καλλιεργειών ε, ε από επικονιάζονται λοιπόν από τις μέλισσε. Δηλαδή αν δεν υπάρχουν πια μέλισσε, δεν υπάρχουν πια καλλιέργειες. Τουλάχιστον δεν υπάρχουν καρποί όπως ε, ε, τα σιτηρά, τα, τα φρούτα, η λίανθη. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος ε, και η ΕΦΣΑ εδώ και μία εβδομάδα στις 16 Ιανουαρίου ε, δημοσίευσε τρεις σημαντικές νομοδοτήσεις ε, για τα τρία νέα νοικοτενοειδή. Θα τις έχετε φαντάζομαι αυτές τις νομοδοτήσεις. Είδατε στα συμπεράσματα ότι στα αγγλικά λέει high acute risk. Ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος τοξικότητας, που είναι σημαντική ένδειξη των επιστημόνων της ΕΦΣΑ που μας ε, προειδοποιεί εμείς ως διαχειριστές του κινδύνου να κάνουμε κάτι, γιατί είναι τρεις από τα πέντε ζυζανιοκτώνα που επιτρέπονται στην οικογένεια των νέων οικοτινοειδών αλλά τρεις από αυτές τις ουσίες έχουν, ενέχουν υψηλό ε, κίνδυνο τοξικότητας για τις μέλισσες. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πώς ε, μπορούμε να μεταφράσουμε στην ε, νομοθεσία αυτές τις τρεις νομοθετήσεις, ε, που είναι πολύ σοβαρές όπως σας υπενθύμησα και προηγουμένως. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε διαδικασία περισσολογής, αλλά πολύ σύντομα η Επιτροπή θα επανέλθει με προτάσεις για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στην νομοθεσία αυτές τις τρεις ε, επιστημονικές νομοδοτήσεις. Αφενός, έχουμε μια μεγάλη μερίδα επιστημόνων ε, που αναγνωρίζουν αυτή την ε, ή μάλλον φορέων, ε, μεγάλη ομάδα φορέων ε, που στηρίζουν αυτές τις νομοδοτήσει. Από την άλλη βεβαίω ε, δεν αποτελεί έκπληξη, έχουμε την βιομηχανία των ζανιοκτώνων, των σπόρων και τους γεωργού που μας λένε προσοχή, αν απαγορεύσετε αυτά τα νέα νοικοτενοειδή που χρησιμοποιούνται κατά κόρον, αυτό θα έχει οικονομικές επιπτώσεις και μάλιστα σημαντικέ ε, Τα στοιχεία που ανέφεραν, εντάξει δεν τα αναλαμβάνω εγώ, εκείνοι τα είπαν, 17 δισεκατομμύρια μέσα στα 5 ε, χρόνια και 50.000 θέσει εργασία στα 5 χρόνια που τίθεται σε κίνδυνο αν υπάρξει απαγόρευση. Από την άλλη, η ανάλυση μας δείχνει ότι η επεξεργασία των ε, σπόρων που ψεκάζονται με ένα ζυζανιοκτόνο, συστημικό ζυζανιοκτόνο, δηλαδή περνάει μέσα από το φυτό και φτάνει στο άνθος για να προστατεύσει το φυτό από ε, τα ζυζάνια. Η επεξεργασία λοιπόν ε, ε, του σπόρου είναι καινοτόμος γιατί δίνει χρόνο στον γεωργό, εξοικονομεί δηλαδή χρόνο γιατί γίνεται πολύ πιο εύκολη είναι η όλη διαδικασία από το τρακτέρ. Και έτσι θεωρούμε ότι είναι μια καινοτόμα μέθοδος που έχει ωφέλη σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο από το τρακτέρ που ψεκάζει ε, ζανιοκτόνο πάνω στα άνθη. Από τις μελέτες όμως ε, φάνηκε ότι αυτά τα νεονικοτενοειδή έχουν τρία αρνητικά στοιχεία. Το πρώτο είναι δηλαδή κατά τη χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή με, με, μέσω σπόρων ή μέσω σπρέι, με οποιοδήποτε τρόπο και αν εφαρμόζονται, υπάρχει ε, η παρουσία του στο νέκταρ. Η παρουσία τους επίσης κατά την ε, μετάβαση του αραβοσίτου που και οι μέλισσες παίρνουν ε, αυτή την υγρασία του αραβοσίτου ως ε, πηγή υγρασίας και τρίτον είναι η σκόνη που απελευθερώνεται όταν εφυτεύεται ο σπόρος του ζωνιοκτώνου ο κόκκος αν θέλετε καλύτερα ή αν, ακόμα και όταν ψεκάζεται. Και αυτή η σκόνη μπορεί είτε να μολύνει ε, άλλες ε, καλλιέργειες που είναι γειτονικέ, όπως οι καλλιέργειες κόλζα, ή οι μέλισσες περνάνε από ένα σύννεφο τέτοιες σκόνης και μολύνονται. Δημιουργούνται λοιπόν έτσι πολλά προβλήματα, όμως θεωρούμε ότι ε, αυτή η μέθοδος με τους κόκκους είναι πολύ πιο καινοτόμο σε σχέση με τον παραδοσιακό ε, τρόπο ψεκασμού. Σήμερα δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω στον κύριο Ντέιβις για τις ε, λεπτομέρειες των ε, μέτρων. Θεωρώ όμως ότι πολύ σύντομα ε, και συγκεκριμένα στην αρχή της επόμενης εβδομάδας θα μπορέσει η Επιτροπή να κάνει ε, ανακοινώσεις για αυτά τα μέτρα που θα προταθούν στα κράτη-μέλη για να ψηφιστούν ε, στο πλαίσιο της Επιτροπολογίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τον λόγο ε, στον, ε, στον συγγραφέα ε, της σχετικής παρουσίασης, τον Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας Ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για τα επιστημονικά ευρήματά μας σχετικά με τα αποτελέσματα ε, των νεονικοτοειδών ε, στις μέλισσες. Ε, το Τμήμα Οικονομικής και Επιστημονικής Πολιτικής ζήτησε από, τον οργανισμό στον οποίο ανήκω, τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό της Αυστρίας, να ετοιμάσουμε ένα σημείο μας σχετικά με τα αποτελέσματα των νεονικοτοειδών στα, στις και το σημείο αυτό δημοσιεύθηκε πέρσι τον Δεκέμβριο. Πέρσι τον Δεκέμβριο. Η Μάρκριτ Γκριμ, η Κάτριν Σέντι και ε, εγώ έχουμε συγγράψει μαζί ε, το έγγραφο αυτό. Εγώ λέγομαι Άλλα Ρίχ, είμαι ε, βιολόγος, ασχολούμαι και με την επιστήμη του έδαφος και την χημεία και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι ρηπαντικές ουσίες στο περιβάλλον. Όσον αφορά το ενημερωτικό σημείωμα για τα νεονικοτοειδή ε, και τις μέλισσες, ε, εξετάσαμε τα πρόσφατα δημοσιευμένα επιστημονικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων άρθρων ε, που έχουν να κάνουν με, το, με τα αποτελέσματα των νοικοτοειδών στις μέλισσες. Αναφορές για ζημιές σε μελίσια έχουν αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη. Τα νεονικοτοειδή ε, είναι εντομοκτώνα που χρησιμοποιούνται ε, σε γεωργικά φυτά ε, για να καταπολεμηθούν διάφορες ε, ασθένειες ε, και συνδέονται όλο και περισσότερο με τις ζημίες αυτές. Ιδιαίτερα κάποιες επιστημονικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν πέρσι, τον, πέρσι το φθινόπωρο που είχαν να κάνουν με τις σχεδόν τοξικές ποσότητες νεονικοτοειδών συγκέντρωσε πολύ προσοχή ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση και η Ευρωπαϊκή Κομισιόν ε, ζήτησε περαιτέρω επιστημονικές μελέτες. Η ε, Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κλήθηκε από την Κομισιόν να κάνει μια μελέτη αντικτύπου σχετικά με τα αποτελέσματα των νέων οικοτοειδών στις μέλισσες. Οι εκθέσεις αυτές δημοσιεύτηκαν πριν λίγες μέρες και θα παρουσιαστούν αμέσως μετά. Ε, η επικονίαση αποτελεί σημαντική υπηρεσία στο οικοσύστημα και ε, υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη πάνω από το 80% των καλλιεργιών ε, βασίζονται σε αυτήν. Γι' αυτό βλέπουμε... Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η αύξηση των αριθμών αναφοράς ζημιών στα μελίσια. Τα νεονικοτονοειδή έχουν υψηλή τοξικότητα για όλα τα είδη μελισσών, ε, αυτές που παράγουν, ε, τις, αυτές που τις άγριες ε, και τους πουπουρές. Πέρα από τα, τους κανονικούς τρόπους έκθεσης, ο συστημικός χαρακτήρας τους ε, επιτρέπει να μεταφέρονται σε όλο το φυτό και έτσι ε, εκτίθενται οι μέλισσες. Πρόσφατες δημοσιεύσεις ε, δείχνουν ότι ακόμα και χαμηλές δόσεις επηρεάζουν την υγεία των, φυτο... των μελισσών. Έχουμε δει τις σχεδόν θανατηφόρες δόσεις στις μέλισσες, οι οποίες οδηγούν σε ε, διάφορες διαταραχές ε, όσον αφορά ε, την, τη μνήμη τους, την ικανότητα να μαθαίνουν κλπ. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι η χρόνια έκθεση σε χαμηλές ε, δόσεις νεονικοτοειδών μπορούν να μειώσουν την ε, δυνατότητα αναπαραγωγής ε, των μελισσών και να οδηγήσουν σε, και να μειώσουν την αντίσταση στις ασθένειες. Επίσης, τα νεονικοτοειδοί μπορούν να οδηγήσουν στη θνησιμότητα ακόμα και σε χαμηλές δόσεις ε, κάνοντας, ε, τις, ε, κάνοντας τα μελίσια πιο ευάλωτα σε, άλλ, σε άλλες διαταραχές. ενώ τα, οι, επιστημονικές μελέτες υπολογίζουν τα μη θανατηφόρα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα έχουν αμφισβητηθεί. Και για να εξετάσουμε πλήρως ε, τον κίνδυνο για τις μέλισσες είναι απαραίτητο να γίνουν ε, περαιτέρω μελέτες ε, που να είναι σχεδιασμένες σωστά και που να διαρκούν αρκετές, αρκετό χρόνο. Μέχρι τώρα κάποιες ε, ευρωπαϊκές χώρες έχουν εφαρμόσει μέτρα τα οποία στόχο έχουν να μειώσουν τις αρνητικές ε, συνέπειες των ε, νέων οικοτονιδών για τις μέλισσες. Ωστόσο, τα μέτρα μείωσης του κινδύνου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο επικεντρώνονται στο να μειώσουν τον κίνδυνο οξίας δηλητηρίασης των μελισσών και δεν, δεν εξετάζουν καθόλου τον κίνδυνο από την χρόνια έκθεση. Όσο, υπάρχουν, ε, ε, όσο υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τα αποτελέσματα των νεονικοτοειδών ε, στις μέλισσες, θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξης κατά την διαδικασία διοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόσωπος της ΕΦΣΑ. Να πω λίγα λόγια και εγώ για τα συμπεράσματα μας ε, για το ίδιο θέμα. Λάβαμε μία εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε και το έργο μας. Ορίζοντας ποιες είναι οι ουσίες που πρέπει να εξετάζουμε, δηλαδή τις ε, νεονικοτιδές ουσίες. 31 Δεκεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκε αυτή η έκθεση και Υιοθετήθηκαν έγκαιρα τα συμπεράσματα και δημοσιεύτηκαν λίγες εβδομάδες μετά. Η Κομισιόν μας ξεκαθάρισε ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις συγκεκριμένες χρήσεις εντός της Ένωσης ε, και σε παιδοσπόρων και κόκκων. Εμείς έπρεπε να λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία κατά τη μελέτη ε, αντικτύπου. Είναι τα δεδομένα λοιπόν των ετούντων που λέμε υπόψη. Των ετούντων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για, ε, δηλαδή ε, καθώς υπέβαλαν την ενεργοουσία, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, ε, με τις άδειε που δίνουν στα προϊόντα φυτοπροστασίας. Λάβουμε υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση ε, για θέματα φυτοπροστασίας εν προκειμένου, καθώς επαναλαμβάνω αυτό το έγγραφο, ένα έγγραφο της ΕΦΣΑ, από το πάνελ της ΕΦΣΑ και είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε για να καταλήξουμε τελικά στο μέλλον σαν έναν οδηγό ε, σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα διωτηθούν ως τα τέλη του Μάη. Λάβουμε υπόψη και άλλες μελέτες, έρευνες, monitoring που έχει γίνει ε, ακριβώς για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Πώς κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα, σύλλαξαμε δεδομένα. Ε, τα στοιχεία που δίνουν οι ετούντες, πληροφορίες σχετικά με τις ε, ε, εγκρίσεις που έχουν και τις άδειες που έχουν δει στα κράτη-μέλη και μετά κάναμε μια αξιολόγηση αυτών των δεδομένων. Θέλω να επισημάνω εδώ ότι το προσωπικό της ΕΦΣΑ έκανε την αξιολόγηση αυτών των δεδομένων. Δηλαδή, δεν χρησιμοποίησαμε ένα πάνελ εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, αλλά η ίδια η ΕΦΣΑ, η υπάλληλη της έκανε την αξιολόγηση. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρω και πάλι την επιστημονική αυτή γνώμη που βασί... πάνω στην οποία βασίζονται αυτά τα προϊόντα φυτοπροστασίας εν προκειμένου. Για να το κάνουμε αυτό, στην αξιολόγησή μας συμπεριλάβαμε όλα τα νέα επιστημονικά στοιχεία και πορίσματα, ιδίως ό,τι αφορά το πώς επηρεάζεται η συμπεριφορά των μελισσών και των κοινότητων τους. και χρησιμοποίησαμε την πλέον σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία προκειμένα. Κάναμε λοιπόν μια μελέτη αντικτύπου με βάση αυτά τα στοιχεία ε, και για τα οξέα συμπτώματα αλλά και τα χρόνια ε, σχεδόν θανατηφόρα συμπτώματα. και ε, που προκαλούνται από τους σπόρους και από κόκκους. Αυτό γίνεται κυρίως με την έκθεση σκόνη όταν ε, γίνεται χρήση και επεξεργασία ε, των σπόρων ή των κόκκων, έκθεση σε υγρά και έκθεση ε, στα εντομοκτώνα και στα υπολείμματα καλλιεργιών. Εκεί δεν είχαμε πάρα πολλά στοιχεία για να καταλήξουμε σε πολύ ασφαλή συμπεράσματα καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα για όλες τις κατηγορίες των ορικοτοδών που εξετάσαμε και τα διαθέσαμε στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το επόμενο βήμα ήταν να κάνουμε μια διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, κυβερνητικούς εμπειρογνώμονες, δηλαδή αυτούς που διόρισαν οι εθνικές αρχές για να ανταλλάξουμε απόψεις με βάση αυτά τα συμπεράσματα. Και μετά καταλήξαμε στα τελικά συμπεράσματα που είναι τα συμπεράσματα, αναλαμβάνω του προσωπικού της ΕΦΣΑ ως ανεξάρτητου επιστημονικού οργανισμού. Ποια είναι αυτά τα κύρια συμπεράσματα. Περίπλοκα είναι. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τα συμπεράσματα σε πίνακες, επισκοπικούς πίνακες, που αφορούν όλους τους χρήστες και απευθυνόμαστε σε όλους τους χρήστες, δίνοντας τα συμπεράσματα για όλες τις πηγές έκθεσης όπως ανέφερα πριν, ε, και εκεί που θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε ε, οξέα και χρόνια συμπτώματα, όπως ανέφερα πριν. Εκεί τουλάχιστον όπου μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα, γιατί είχαμε αρκετά δεδομένα. Επίσης, τα αποτελέσματα αξιολόγησης οδήγησαν στο ότι, όπως είπα, επειδή υπήρχε ένα και δεδομένων, δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις υπήρχαν αρκετά δεδομένα και καταλήξαμε σε συμπεράσματα. Έπειτα, σε άλλες περιπτώσεις, μπορούσαμε με να κάνουμε μελέτη αντικτύπου, αλλά δεν εντοπίσαμε κίνδυνο για μία συγκεκριμένη καλλιέργεια και μία συγκεκριμένη ε, οδό έκθεσης σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαμε διαθέσιμα δεδομένα για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη κινδύνου. Ε, παράδειγμα, δεν είχαμε επαρκή στοιχεία για την ε, έκκληση σκόνης για, από όλες τις πηγές. Όπως δεν είχαμε όλες τις πληροφορίες και τη συγκέντρωση σε νέκταρ και γύρι. Είχαμε στοιχεία για κάποιες καλλιέργειες αλλά όχι για όλες. Επίσης δεν είχαμε επαρκή στοιχεία σε ό,τι ε, αφορά την ε, συχνότητα ε, της επικονίασης και στα ρευστά, στα υγρά, συγγνώμη, εν Προσπαθήσαμε να κάνουμε ως έναν κατάλογο, όσο γίνεται πιο ξεκάθαρο, όλα τα στοιχεία και πού είναι επαρκή τα στοιχεία και πού είναι λυπή τα στοιχεία. Τώρα να επανέλθω στι κύριε μεθόδου μεθόδους έκθεσης, βάσει των οποίων μας ζητήθηκε αυτή η μελέτη ε, και η ανάλυση κινδύνου. Μπορώ να συνοψίσω το αποτελέσμα ω εξή. Η έκθεση στο Ινεγύρι και το Νέκταρ, συμπέρασμα, μόνο οι χρήστες ε, μπορούν να θεωρηθούν ότι μπορούν να έχουν ένα χαμηλό κίνδυνο. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι καλλιέργειες που προσελκύουν μέλισσες, είτε θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη που να υποδεικνύει κάποιο κίνδυνο ή δεν έχουμε παρκή στοιχεία για να καταλήξουμε σε μία ε, αξιόπιστη ε, μελέτη. Δεύτερον, η έκθεση στη σκόνη. Ο κίνδυνος για τις μέλισσες ήταν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί με κάποιες εξαιρέσεις όπως η χρήση στα σαχαρότευκλα όπου υπάρχει η συγκεκριμένη περίπτωση Επεξεργασία ε, σπόρων, που είναι ειδική διαδικασία για τα ζαχαρότευτλα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θεωρήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι την έκκληση σκόνης, όπως επίσης και για τις καλλιέργειες σε θερμοκήπια και τη χρήση κάποιων κόκκων. Εκεί θεωρήσαμε ότι ο, ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Τέλος. Και τέλος άλλες μορφές έκθεσης ε, δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αξιόπιστα δεδομένα. Για παράδειγμα, έχουμε την περίπτωση της επεξεργασίας ε, αραβόσιτου, ε, όπου εκεί είδαμε ότι μπορεί να καταδεχθεί ένα επίπεδο ε, κινδύνου. Παρόμοια συμπεράσματα για ένα τέταρτο εντομοκτόνο που δεν είναι νεονικοτοειδές, αλλά είναι το φιμπρονίλ, ε, το οποίο είναι, έχει παρόμοια χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία θα σας τα δώσουμε στα τέλη Μαρτίου. Ευχαριστώ πολύ. Να ε, ξεκινήσουμε από τον Κρίς Ντέιβις. Παρακαλώ, Κρίς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναβάλαμε την ε, συζήτηση αυτή για να ακούσουμε τα, έστω και προσωρινά αποτελέσματα της ε, ΕΦΣΑ ε, και χαίρομαι που το κάναμε διότι ήταν πολύτιμη η παρέμβαση. Αν και αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με το ότι ο κόσμος πιστεύει ότι οι μέλισσες είναι πολύτιμες για μας, όχι μόνο λόγω ε, του ρόλου τους ε, στην ε, ε, επικονίαση. Είναι περίεργο διότι γενικά δεν είναι πολύ δημοφιλή τα έντομα εκτός από τις μέλισσες και τις πεταλούδες. Ότι Γράφει εδώ ότι ο περιορισμός των νεονικοτοειδών λόγω των δυνάμει κινδύνων δεν θα κάνει τίποτα για να βελτιώσει τη γενική υγεία των μελισσών. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κάποιος να κάνει μια τέτοια ε, δήλωση δεδομένων των ε, στοιχείων που ακούσαμε. Αυτό φαίνεται να είναι λάθος. Ε, δεν πιστεύω και... Νομίζω ότι είναι σαφή τα στοιχεία κατά των νέων Ε, Στην καλύτερη περίπτωση είναι σχεδόν θανατηφόρα η επίδρασή τους. και οι συνέπειες αυτές οδηγούν ε, σε ε, ε, λιγότερη αντίσταση στις ασθένειες και σε χαμηλότερη δυνατότητα αναπαραγωγής. Αυτό δεν είναι νέο. Διάφορες εθνικές κυβερνήσεις το εξετάζουν αυτό εδώ και 15-16 χρόνια νομίζω. Νομίζω ότι η γαλλική κυβέρνηση εισήγαγε απαγόρευση για κάποια φάρμακα, ένα της Μπάγερ το 1999, και κάποια φάρμακα για το ε, καλαμπόκι το 2004. Κάποια, κάποιες εθνικές κυβερνήσεις λοιπόν ενήργησαν με βάση τις, ε, τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους και χρησιμοποιώντας την αρχή της προφύλαξης. Ε, ο βιομηχανικός ε, τομέας των φυτοφαρμάκων θα πει ότι υπήρξαν τεράστιες απώλειες στη, στην σχετική βιομηχανία και αναγνωρίζω ότι ε, τα φυτοφάρμακα ε, έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο, ε, αλλά θα πρέπει να βασιστούμε στα επιστημονικά στοιχεία και να λάβουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα και να ενεργήσουμε ανάλογα. Ο σχετικός βιομηχανικός τομέας θα πει ότι η απογόρευση οδηγεί σε τεράστιες ζημιές, αλλά ε, κοίταξα την ε, μελέτη τη της περιβαλλοντικής υπηρεσίας ε, που αν δεν έχει δημοσιευτεί θα δημοσιευτεί σύντομα. Εμένα κάποιος από την Κοπεχάγη μου στείλε ένα αντίτυπο Ε, εάν κοιτάξει λοιπόν ε, στην Γαλλία το αποτέλεσμα της απαγόρευσης βλέπουμε ότι στην παραγωγή δεν είχε σχεδόν καμία συνέπεια και μάλιστα ε, η καλύτερη χρονιά ήταν κάποια χρόνια μετά την απαγόρευση του συγκεκριμένου προϊόντος για το καλαμπόκι. Πάντως ε, αναγνωρίζω ότι ε, τα φυτοφάρμακα έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο, αλλά η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι μέλισσες δεν έρχονται σε επαφή με τα φυτοφάρμακα αυτά. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει αυτό. Σε κάποια μέρη θα πρέπει να ε, εισάγουμε περιορισμούς ή απαγορεύσεις όσον αφορά τη χρήση κάποιων προϊόντων για κάποιες καλλιέργειες τις ε, καλλιέργειες που προσελκύουν περισσότερο τις μέλισσες. Σε άλλες περιπτώσεις, ε, ίσως πρέπει να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές, όπως ήδη έχουμε σε κάποιους τομείς, ε, να, ε, να περιορίσουμε, για παράδειγμα, ε, τον ψεκασμό. Ε, να απαγορεύσουμε για παράδειγμα τον ψεκασμό ε, νεονικοτοειδών πάνω σε, σε ε, ανθοφόρα φυτά. Η Κομισιόν είπε, μήπως μπορείτε να το αυτό, είπε ότι πολύ σύντομα και μπορεί να τα πείτε στο Συμβούλιο αντί για το Κοινοβούλιο, αλλά είπατε ότι ε, πολύ σύντομα θα υποβάλλετε συγκεκριμένε προτάσει. Τι φύση θα έχουν αυτέ οι προτάσει, ε, θα προτείνετε ε, νομοθετικά μέτρα ή απλά θα προτείνετε την ε, εισαγωγή κατευθυντηρίων γραμμών και περαιτέρω μελέτε. Ευχαριστώ πολύ και άλλοι έχουν ζητήσει το λόγο. Η Κρίστα Κλάς. ζητησει το λογο η κριστα Κλά. ευχαριστω Προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Μόλις μιλήσαμε για μέλη, ακούσαμε πολύ καλές εξηγήσει από ε, την Κομισιόν και το σημαντικό είναι και το ανέφερε ο, ε, ε, ο χρειαζόμαστε τις μέλισσες όχι μόνο για την παραγωγή μελιού, αλλά χρειαζόμαστε και για την επικονίαση των φυτών. Πρέπει να τα προστατεύσουμε λοιπόν. Ε, και θα πρέπει ε, να το δούμε αυτό ε, και πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να δούμε και τα φυτοφάρμακα τα οποία προστατεύουν τα, φάρμακα, τα φυτά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και τη διάσταση αυτή. Είναι πάρα πολύ ανησυχητική η κατάσταση και αν εφαρμόσουμε την Ε, αρχή της ε, προφύλαξης, ε, τότε ήδη έχουμε καθυστερήσει, διαπιστώνουμε όταν διαβάζουμε τη μελέτη αυτή. Εάν αναφέρεται εδώ η τοξικότητα. Θα πρέπει να εξετάσουμε την βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων από ό,τι άκουσα έχουν ληφθεί και τα δύο υπόψη κατά την εξέταση του θέματος. Ε, το θέμα είναι όμως ότι εδώ πρόκειται για ένα σημαντικό ε, όπλο για την φυτοπροστασία που ε, που το χρειαζόμαστε απαραίτητα. Ε, υπάρχουν ε, κάποιοι ε, γεωργοί που δεν ψεκάζουν κάθε χρόνο τα φυτά τους, λαμβάνοντας υπόψη και τους σχετικούς κινδύνους. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι παράγοντες εδώ που πρέπει να ληφθούν υπόψη, γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Τι εναλλακτικέ μέθοδοι υπάρχουν και μας είπατε ότι η Γαλλία ήδη έχει μια απαγόρευση για το καλαμπόκι. Στη Σλοβενία υπάρχει μερική απαγόρευση, εξετάστηκε εκεί μήπως ε, οι μέλισσες ε, τα πάνε καλύτερα, διότι ε, μας ενδιαφέρει και αυτό πώς θα λειτουργήσει τελικά μια απαγόρευση. Και τι μπορεί να κάνει κανείς ε, αμέσως, διότι υπάρχει τώρα, εδώ και τώρα, διότι υπάρχει μια υποψία. Και βλέπουμε ότι με λάθος ε, χρήση γίνονται πράγματα τα οποία δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει εδώ και τώρα να λάβει μέτρα και εγώ σκέφτομαι πιο πολύ τη βιώσιμη χρήση. Ε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ε, πιο αυστηρό έλεγχο και να επιτρέψουμε σε κάποιες ειδικέ περιπτώσεις τη χρήση. Θα πρέπει λοιπόν προληπτικά να ε, προωθήσουμε την ε, βιώσιμη χρήση των ε, φυτοφαρμάκων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Στάνθος Πελιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε αυτή τη συζήτηση εδώ σήμερα. Χαίρομαι που, αν και έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρεις ημέρες αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή Αναφορών, ξεκινάμε όμως και με τη συζήτηση και με την Επιτροπή που μας ε, ε, έδωσε κάποιες απαντήσεις και τότε και σήμερα σε ό,τι αφορά τις τελευταίες μελέτες ε, της ΕΦΣΑ είναι κάτι που μας καθησυχάζει ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά την εξολόγηση των ε, κινδύνων και των επιστημονικών επιχειρημάτων. Θέλουμε να δούμε ποια είναι η δράση που μπορούμε να αναλάβουμε. Υπάρχουν εμπόδια γιατί το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η Επιστημονικέ αξιολογήσεις δεν είναι καινούργιε ούτε αυτές. Η συζήτηση ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξαναγίνει και η τελευταία έκθεση στην οποία κληθήκαμε να πάρουμε, να πάρουμε θέση ήταν το 2011 για ένα σχέδιο ε, πάλης ε, κατά της θρησιμότητας των μελισσών. Επομένως, ως με τους οικολόγους μπορούμε να πούμε δυστυχώς ότι δεν πήγε ε, αρκετά μακριά. Πρώτα απ' όλα στα ζυζανιοκτώνα και την τοξικότητά τους. Ε, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τα πιο ε, ζημιογόνα ζυζανιοκτώνα για τις μέλισσες και συγκεκριμένα για τα νεονικοτενοειδή, για τα γενικά τροποποιημένα και ούτω καθεξής. Ε, ε, εξακολουθεί να ισχύει η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει και η αρχή της πρόληψης. Δεν θα, θα επιστρέψω στην προηγούμενη συζήτηση για την ε, οδηγία για το μέλι. Και τέλος, ένα από τα επιχειρήματα που... που έχουν θυγεί και στο παρελθόν, τα γενικά οικολογικά προβλήματα που συνδέονται με τη μονοκαλλιέργεια και σημαίνουν και την ανάγκη πιο βιώσιμων ε, μεθόδων και πρακτικών. Ήδη το 2011 είχαμε κάνει μια τέτοια συζήτηση. Ε, είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει η σύνδεση μεταξύ της θνησιμότητας ε, των μελισσών και των ζωνιοκτώνων και ίδιο στοιχείο προβληματισμού σε ό,τι αφορά την σύνδεση μεταξύ των γενικά τροποποιημένων οργανισμών και τη θεσιμότητα των μελισσών. Ήταν ένα από τα επιχειρήματα που ε, αιτιολογούσαν την αδράνεια. Τέλος, 2012, τρει μελέτες και πλέον φτάνουμε στο 2013 για τα γάματα φαομικρών θα τα ξανασυζητήσουμε, για τα ζυζανιοκτώνα από την προηγούμενη εβδομάδα στηριζόμαστε στην γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Ο κίνδυνος έχει, είναι πλέον αποδεκτός. Υπάρχει και επιστημονικά πλέον αυτή η σύνδεση μεταξύ των ζυζανιοκτώνων και, και της θνησιμότητας. Περιμένουμε και μια πληρέστερη έκθεση στα τέλη 2013. Επομένω, πλέον δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για την απαγόρευση τη θέση εμπορία των συζανιοκτών αυτών στην ευρωπαϊκή αγορά. Ε, υπάρχουν και αναφορές όπως σας είπα από τους ε, πολίτε, Οι δύο αναφορές ε, που εξέτασε η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου την τελευταία εβδομάδα αφορούν πάνω από 80 οργανώσει οργανώσεις που απευθύνθηκαν σε εμά. Η μία αναφορά αφορούσε την υιοθέτηση μέτρων για την απαγόρευση ορισμένους ζανεοκτώνων που επηρεάζουν και την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των μελισσών. Και η δεύτερη αναφορά αφορούσε τη σύνδεση με την χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Και σήμερα στο ημικύκλο θα είδατε ότι υπάρχουν 1.250.000 πολίτες που μας ζητούν να πάρουμε μέτρα για να ε, καταργηθεί ένας από τους βασικούς ε, κινδύνους και τις απειλές για τις μέλησες Θα ε, απευθυνθούν λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε μερικές μέρες για να δράσει αυτή να τον πιο σύντομα. Και σε επιστημονικό επίπεδο και στην ανάγκη ανταπόκρισης στους πολίτες μας μπορούμε σήμερα να πάρουμε μέτρα για να θέσουμε τέλος σε μια οικολογική, περιβαλλοντική αλλά και οικονομική καταστροφή. Οι παραγωγοί ζενοκτώνων λένε ότι θα έχουμε τεράστιε ε, ε, απώλειες οικονομικές. Εντάξει, υπάρχει εδώ πέρα μια πάλι αριθμητικών στοιχείων. Εμεί έχουμε αντίθετα στοιχεία που λέμε ότι με, τη, με αυτή την πολιτική που προτείνουμε θα δημιουργηθούν 1,2 εκατομμύρια θέσει εργασία. 17 δισεκατομμύρια απώλειες. Ε, ποιο είναι το οικονομικό ε, κόστος που συνδέεται με το κόστος ε, των μέλισσών που αν σκεφτείτε σε τελική ανάλυση η επικονίαση είναι μια δωρεάν υπηρεσία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το στάδιο η απόφαση είναι απλώς πολιτική. Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα, ε, δυσκολεύεται η Επιτροπή να ε, αναλάβει δράση ε, σύντομα για την απαγόρευση της χρήσης των νεονικοτενοειδών μέσα στο άμεσο μέλλον. Ελπίζω οι πολίτες να μπορούν να βασιστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είμαστε πιο φιλόδοξοι στα μέσα που έχουμε σε σχέση με τις ψηφοφορίες μας πριν από δύο χρόνια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πραγματικά είναι πορεία άξιο πώς <clears throat> εγκρίθηκαν αυτές οι αυτά τα φυτοφάρμακα στην αρχή. Ε, και αποτελεί σίγουρα ένα χτύπημα στην αξιοπιστία του συστήματος έγκρισης στην, ε, στην Ευρώπη. Η, το θέμα των νοικοτινοειδών βέβαια πέρα από τι λέγανε οι επίσημες αρχές ευρωπαϊκές <clears throat> για τους πολίτες της Ευρώπης ήταν ξεκάθαρο. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι η τρίτη σε παραγωγή με πανευρωπαϊκά, 17η στον κόσμο. Οι, μελισσοκόμοι μας αντιμετωπίζανε ε, το πρόβλημα της επιπτώσης των νοικοτινοειδών χρονιά με τη χρονιά, με πολλούς θανάτους μελισσών <clears throat> και αυτό επειδή και η μια άλλη αιτία των θανάτων αυτών είναι και οι μεταλλαγμένες καλλιέργειες αξίζει να δούμε αν η Επιτροπή και η ΕΦΣΑ θα ε, επαρεξετάσει τη θέση της και για τα μεταλλαγμένα. Ε, σε κάθε περίπτωση είναι σαφέστατο ότι πρέπει οπωσδήποτε να ε, προχωρήσουμε στην απαγόρευση αυτών των ουσιών. Το κόστος για την κοινωνία μας και για, τις, και για, το, για τις κλάδους αλλά και για την κοινωνία μας μέσα από την γεωργική παραγωγή και την κατάρρευση των επικονιαστών μας θα είναι συγκλονιστικό και περιμένουμε και ζητάμε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε από την Επιτροπή προ αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφο Κόλλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα, το ανέφερε και ο Κρήτον, το πώ δίνονται οι άδειε και το γεγονό ότι περιμένουμε πρώτα να αποδεχτούν οι βλάβε για να αποσυρθούν ε, επικίνδυνα προϊόντα τα οποία έχουν εισαχθεί βέβαια πρώτοι και έχουν χρησιμοποιηθεί. Αλλά δεν ήθελα να ανοίξω τώρα αυτό το θέμα γενικότερα, ήθελα να αναφέρω όμω ε, κάποιες ιδιαιτερότητες που υπάρχουν τώρα και στην Ελλάδα για τη χρήση των ε, νεονικοτινοειδών. Όπω θα ξέρετε υπάρχει ε, αυτό το κόκκινο καθάρι, το οποίο απειλεί τους φίνικες και έχουν εξεταθεί πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν πολλά περιστατικά στην Ελλάδα που πολίτες είχαν πρόσβαση σε παρόμοια φυτοφάρμακα, τα χρησιμοποίησαν και υπάρχουν μαζικοί θάνατοι μελισσών ε, και ιδιαίτερα σε νησιά, οπότε είναι και ένα επιπλέον παράδοση που θα πρέπει να εξεταστεί, γιατί υπάρχει εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε διάφορα επικίνδυνα σκευάσματα, ε, είτε υπάρχει συνταγή γεωπόνου, είτε δεν υπάρχει και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στην ε, εξέταση επικινδυνότητας και αυτό το παράγοντα ότι σήμερα τα φυτοφάρμακα είναι διαθέσιμα εύκολα στην αγορά και υπάρχει πρόσβαση ανθρώπων που δεν ξέρουν ε, να τα χρησιμοποιούν έστω με κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκέρλινγκ. just um, incompetence. Um, Όχι, εγώ δεν τα κατάφερα μόνο να ανοίξω το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Ε, θα προσπαθήσω να τραβήξω αυτή τη συζήτηση και πάλι στο θέμα το οποίο συζητάμε αυτή την Επιτροπή για όσο καιρό συμμετέχω εγώ σε αυτήν. Δηλαδή, ε, τον αναλογικό αντίκτυπο των νέων νοικοτονοειδών ε, στην υγεία των μελισσών. Έχουμε καταδείξει στη, στην έκθεση μας ε, στο Κοινοβούλιο, γιατί δεν ε, ε, είναι μόνο ένας παράγοντας, μόνο μία η αιτία της εθνισμότητας των μελισσών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι ε, παρασίτων, καιρικών συνθήκων. Όλα αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν. Επομένω, όταν εξετάζουμε τις ε, δοκιμέ και τα αποτελέσματα, πρέπει να εξετάζουμε και αυτά τα ζητήματα των παραγόντων. Δεν πρέπει δηλαδή να, να ε, απαγορεύσουμε απλώ μία από αυτέ, τις να καταργήσουμε μία από αυτέ τι αιτίε. Εγώ χαιρετίζω απολύτω ε, ε, την έκθεση τη ΕΦΣΑ, είναι πρόσδεκτη, απλά δεν πάει αρκετά μακριά, γιατί συζητάμε ξανά και ξανά αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας και περιμέναμε τόσο καιρό και διστάζαμε να κάνουμε κάτι μέχρι να λάβουμε αυτή την έκθεση και αντί να τη συζητήσουμε με ένα λογικό τρόπο, ε, τρέχουμε κατευθείαν προς την απαγόρευση των προϊόντων κατά συνέπεια της έκθεσης, που είναι κάτι δυσανάλογο κατά τη γνώμη μου. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εδώ είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις από πλευράς ε, αξιολόγησης ε, κινδύνου και όπως αναφέρθηκε, χρειάζεται μια εντελώς ε, καινούρια ε, διαδικασία εξελόγησης εκτίμησης κινδύνου. Η διαδικασία λοιπόν τώρα είναι εντελώ διαφορετική από ό,τι ίσχυε στο παρελθόν με άλλα προϊόντα ε, προστασία τη υγεία των φυτών. Επανέρχομαι λοιπόν στο βασικό σημείο για μένα. Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε εδώ είναι κατά τη διαχείριση κινδύνου ε, αναφερόμαστε σε ωφέλη. Ακούσαμε κάποια στοιχεία για τα ωφέλη για τους ε, Ευρωπαίους ε, γεωργούς από την χρήση αυτών των ουσιών. Πρέπει να τα εξετάσουμε πραγματικά ενδελεχώς πριν περάσουμε στην απαγόρευση των προϊόντων. Πρέπει να εκτιμήσουμε και τον κίνδυνο της χρήσης των προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται εδώ και πολύ καιρό είναι σαφές και αναντήρητη αλήθεια ότι τα ζυζανιοκτώνα σκοτώνουν τις μέλισσες. Κανένας δεν το αμφισβητεί. Είναι η μέθοδος ε, με την οποία χρησιμοποιούνται και με την οποία εφαρμόζονται και πρέπει να εξετάσουμε αυτό ενδελεχέστερα. Είχαμε από την ΕΦΣΑ σαφή αποδοχή του γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη δεδομένων, κάτι που επηρεάζει και τα αποτελέσματά του Κάποιες από αυτές τις ελλείψεις ε, αφορούν την εφαρμογή και χρήση. Τα κενά αυτά επίσης συνδέονται και με το γεγονό ότι χρειαζόμαστε περισσότερε επιτόπιε δοκιμέ. Όμω πρέπει να αποδεχθούμε ότι αυτό θα πάρει πολύ καιρό, γιατί επηρεάζονται και από τι καιρικέ συνθήκε. Αν έχουμε 12 μήνε, μπορεί να έχουμε πολύ περίεργε καιρικέ συνθήκε που κάτι που βλέπουμε όλο ένα και πιο συχνά, ε, και φαινόμενα που δεν επαναλαμβάνονται για τα επόμενα 6, 10, 15 χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν αυτή τη στιγμή να πω ότι δεν πρέπει οι συνάδελφοι να χρησιμοποιούν τέτοιε διατυπώσει ότι το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή ξεκάθαρα να, ε, να απαγορεύσει αυτά τα ζωνιοκτώνα. Όχι, καθόλου δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Ε, δέχομαι ότι κάποιοι ε, θέλουν να ακολουθήσουμε αυτή την οδό και εγώ σέβομαι το δικαίωμά σα να το λέτε, αλλά δεν είναι η φωνή του Κοινοβουλίου, δεν είναι κάτι που έχει ψηφιστεί και συμφωνηθεί. Επομένω, μην χρησιμοποιείτε τέτοιε εκφράσει, παρακαλώ, γιατί είναι παραπλανητικέ. είναι κάτι που με φαίνει σε δύσκολη θέση. Γιατί εξορισμού, αν κάποιο είναι υπέρ των βιολογικών προϊόντων, δεν ε, συμφωνεί με τη χρήση ζανιοκτώνων. Αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Δεν εκπλήσουμε λοιπόν που ε, εκφράζεστε έτσι, αλλά δεν είμαστε όλοι στην ίδια θέση. Και ως Επιτροπή θα έπρεπε να συνομιλούμε με την ΕΦΣΑ για να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ε, κατάλληλη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου για να διασφαλίσουμε ότι ο, ο τρόπος χρήσης των προϊόντων αυτών μετριάζει του κινδύνου. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει σε σημαντικό βαθμό. Τέλος, να πω ότι ε, πολύ λυπάμαι που η Επιτροπή λέει ότι θα, θα δημοσιεύσει κάτι την επόμενη εβδομάδα όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα και υπάρχει στην ημερήσια διάταξη εδώ και πολύ καιρό. Ε, θα ήταν είναι πολύ κρίμα που δεν έχουμε έστω κάποιες ενδείξει για το τι θα ήταν ε, αυτή η δημοσίευση. Ε, θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα και δεν θα καταλήγαμε στο ίδιο διέξοδο που θα φτάσουμε σήμερα. Θα πρέπει να το ξαναφέρουμε στην ημερήσια διάταξη που βεβαίω θα το κάνουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ κυρία Κέρνιγκ. Ο Αντρέα Ακούσαμε σήμερα ότι πιθανότατα υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη θνησιμότητα στις μέλισσες και τα χημικά αυτά προϊόντα. Στα νεονικοτινοειδή. Η Κομισιόν είπε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα μελετάει το θέμα. Θα πρέπει να δούμε τι έχει να μας προτείνει. Άλλωστε, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες ε, είπαν σαφώς ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε την ε, αρχή της προφύλαξης. Έχουμε σαφή στοιχεία από τους εμπειρογνώμονες και θα πρέπει να λάβουμε σχετικές αποφάσεις. Ας υποθέσουμε μάλλον ε, νομίζω ότι εμείς οι Ιταλοί βρισκόμαστε στην ε, ε, εμπροστοφυλακή στα θέματα αυτά. Έχουμε εφαρμόσει σταδιακή μείωση και απαγόρευση των νεονικοτοειδών για το καλαμπόκι. Πολλοί μίλησαν για αρνητικές συνέπειες ε, στη γεωργία, εμείς δεν είδαμε καμία πτώση στην ε, παραγωγή του καλαμποκιού, για παράδειγμα. Ίσως λοιπόν μπορείτε να θεωρήσετε την Ιταλία σαν εργαστήριο, σαν ε, πείραμα. Εδώ και αρκετό καιρό δεν χρησιμοποιούμε τα νεονικοτοειδή. Νομίζω θα, θα μπορούσατε να μας θεωρήσετε παράδειγμα. σε κάποιες μέλισσες ε, το ποσοστό θνησιμότητας είχε αυξηθεί στο 50% ενώ τώρα έχει εξαφανιστεί τελείως ε, και φαίνεται να είναι απόλυτα υγιεί οι μέλισσες μας ε, παρότι βέβαια πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες. Νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξη Να μην ξεχνάμε ότι πέρσι τον Απρίλιο, το 2012 δηλαδή, εδώ στο Κοινοβούλιο υιοθετήσαμε έκθεση για την βιοπικιλότητα πρέπει να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα. Οι μέλισσες ε, όλων των ειδών μπορούν να ε, βλαφθούν από ε, τις ουσίες αυτές. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να υιοθετήσουμε κάποια μέτρα. Η Κομισιόν μίλησε για την βιομηχανία των φυτοφαρμάκων, η οποία ανησυχεί πολύ σωστά. ανησυχεί ότι μπορεί να χαθούν θέσεις εργασίας, μείωση του κέρδους. Αλλά, καθότι το 80% των καλλιεργιών απαιτούν ε, έντομα για την επικονίαση, εάν διατηρήσουμε το status quo, ποιο θα είναι αυτό το κόστος για τη γεωργία. Πιστεύω λοιπόν ότι τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Πρέπει να εφαρμόσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες που λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξης. Ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα κανένα, διότι έχουμε ακόμα λίγο χώρο στον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπούμε ιδιαίτερο αλλά συμφωνώ με την κυρία Κέρλ. Δεν ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζήτησε απαγόρευση των νοικοτηδών στην Ευρώπη. Μόνο η Επιτροπή μας. Μόνο στην Επιτροπή α, και στην Επιτροπή Γεωργίας χάσαμε την ψήφο. Μόνο 170 συνάδελφοι μας στήριξαν σε αυτή την έκκληση για απαγόρευση. Λοιπόν, με ιδιαίτερο και το λέω δημοσίω. Πριν από ένα χρόνο είχα και εγώ υποβάλει ένα παρόμοιο ερώτημα στην Κομισιόν. Σαν αυτή την ερώτηση του Chris Davis. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω μια αλλαγή στάσης. Γιατί τότε ξέρετε τι είχε απαντήσει η Κομισιόν έως σήμερα δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα παραστοκτόνα φυτοφάρμακα με τα ναρκωτιδή και δεν μπορεί κανείς να, να πει ότι θεσπίζεται τέτοια σχέση. Χαίρομαι ιδιαίτερα με αυτή τη μεταστροφή της Κομισιόν. Παραμένουν όμως ε, πολλά ερωτήματα. Δεν είναι σαφής ο ορισμός του harmful effect. Τι είναι αυτή η επιβλαβής ε, επιρροή. Ξέρετε, χρησιμοποιούμε όρους που είναι ευέλικτοι και ευπροσάρμοστε, αλλά πρέπει να ορίσουμε ακριβώς τι εννοούμε με αυτό το harmful effect. Η εύσα λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ε, οι μέλισσες είναι ένα πραγματικά περίπλοκο είδος. Δεν μας αφορά μόνο η άμεση τοξικότητα στους ανθρώπους, αλλά και πώς επηρεάζουν γενικότερα το περιβάλλον. Είναι ένα κοινωνικό ε, έντομο η μέλισσα. Και ακόμα και αν δεν υπάρχει άμεση τοξικότητα στον άνθρωπο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα για την κοινότητα των μελισσών. Η Κομισιόν λέει ότι εφάρμοσε μέτρα άμβλυνσης. Πώς μπορεί όμως να ελέγξει την εφαρμογή αυτών των μέτρων όταν ιδίω μιλάμε για μέτρα με σκοπό τη μείωση της τοξικής ε, σκόνης ε, συγκεκριμένων σπόρων. Και βασίζεται η Κομισιόν στα στοιχεία που δίνει η βιομηχανία. Εντάξει, οι ενεξάρτητες ε, μελέτες δεν μπορούν πολλές φορές να βασιστούν σε εξάρτητα στοιχεία. Αλλά όταν λέτε εσείς Κομισιόν εξάρτητες μελέτες, πώς το στηρίζετε αυτό για τη δημόσια υγεία και για την προστασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να κάνουν εξάρτητε μελέτε που να μην λαμβάνουν ε, υπόψη μόνο στοιχεία τη βιομηχανία. Και παραμένει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Σήμερα με τον κανονισμό του 2009, ο 1107, μιλάει για συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δεν έχουμε και γι' αυτό η έφταση σήμερα μιλά για υψηλό κίνδυνο. Δεν βλέπω άλλο μέτρο που θα μπορούσε να προτείνει η Κομισιόν ε, πέρα από την ε, απόσυρση την αγορά όλων των νοικοτήτων. Εγώ θέλω να ακούσω από την Κομισιόν. Θα τα αποσύρει από την αγορά. Ευχαριστώ. Thank you, Pavel. Next speaker, Ευχαριστώ, Μπάρτ Eh, Ευχαριστώ. Δεν θα τα επαναλάβω όλα γιατί έχουν υποθεί. Αν κατάλαβα καλά τα όσα είπαν όσοι προετοίμασαν αυτές τις δύο μελέτες, τι είπαν, ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, αλλά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει υψηλή ε, τοξικότητα, αυτό το ανέφερε και ο συνάδελφος στην Επιτροπή και αυτό που φαίνεται και διαφαίνεται από όλο αυτό το φάκελο ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου. Λοιπόν, προς την Επιτροπή ε, θα υποβάλλετε προτάσεις την επόμενη ε, Δευτέρα στο Συμβούλιο Υπουργών. Κύριε Ποντιλέ, δεν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις τουλάχιστον γιατί υπάρχουν δύο ε, τεινά. Είτε θα μας πείτε συνεχίζουμε με την πεπατημένη, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, να μελετούμε, ε, να χρηματοδοτούμε και ε, θα συνεχίσουμε λοιπόν ε, τον ίδιο δρόμο ή θα δράσουμε με την αρχή της πρόληψης, θα προσαρμόσουμε την κατάσταση, η αδειοδότηση θα σταματήσει η αδειοδότηση αυτών των ε, προϊόντων και βεβαίως και θα συνεχίσουμε με τη μελέτη. Κανένας δεν πρόκειται να σας πει το αντίθετο. Κύριε Πουντλέ, κύριε Μπόρχ, επίτροπε, ε, νομίζω ότι έχετε κάποια μέσα και εργαλεία στα, στη διάθεσή σας για να περάσετε πράγματι σε αυτή την απαγόρευση. Χάρη ε, ε στους συνεργάτες ε, της ομάδας, Έχω εδώ μπροστά μου την ε, ε, νομοθεσία για τα ζανιοκτώνα, ε, εκθέσεις Μπράιερ, γιατί εκείνη ήταν υπεύθυνη των διαπραγματεύσεων και στο παράρτημα 2, σημείο 83, αναφέρεται ρητά ότι εσείς ως Επιτροπή μπορείτε, θα το πω στα αγγλικά καλύτερα, μπορεί να εγκρίνετε λοιπόν μια ενεργός, μια δραστική ουσία μόνο υπό τους προτινόμενους όρους ε, χρήσης ε, των ε, προϊόντων φυτοπροστασίας και με δύο συγκεκριμένους όρους. Ένα, ότι θα οδηγεί σε αμεληταία έκθεση των μελισσών ή δύο, δεν έχει απαράδεκτες χρόνιες και οξύες επιδράσεις στους, στις μέλισσες, ούτε επηρεάζει τη συμπεριφορά τους. Εδώ Θεωρώ λοιπόν κύριε Ποντιλέο ότι έχετε τα μέσα να προτείνετε την επόμενη Δευτέρα ε, την ανάληψη δράσης και πράγματι ε, την απαγόρευση, τουλάχιστον την προσωρινή απαγόρευση των προσωρινών με υψηλή τοξικότητα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράιμερς. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή δείχνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερες γνώσεις ακούω πώς εκπονούνται οι έρευνες και επανειλημμένα με έχει καταπλήξει αυτό. διότι από τη μία επικρίνονται οι έρευνες που, που ανατίθενται από, από τη βιομηχανία σε κάποιον, αλλά και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν είναι πιο αντικειμενικές. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφή εικόνα με τι βάση χρησιμοποιούμε και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις μελέτες για να μπορέσουμε να έχουμε μια, ε, μια επισκόπηση. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ε, απαγορεύσεις ε, βιαστικά. Πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε αποφάσεις ε, σε αντικειμενική βάση και όταν μιλάμε για την έγκριση ή όχι ε, ενός φυτοφαρμάκου, ε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και στα ανθρώπινα φάρμακα υπάρχει ε, στη συσκευασία ένα σημείωμα που μιλάει για τις παρενέργειες, αντενδείξεις κλπ. Δεν μπορούμε να απαγορεύουμε αμέσω οποιοδήποτε προϊόν έχει την ε, παραμικρή ε, παρενέργεια, διότι ε, έτσι καταλήγουμε σε δυσανάλογα μέτρα. και κάτι τέτοιο θα, και θα είχε σημαντικές ε, συνέπειες στη ζωή μας αν είμαστε υπερβολικά αυστηροί. Νομίζω ότι πρέπει να ζυγίσουμε σε ποιες ισορροπίες δικαιολογείται, σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται μια απαγορεύση και σε ποιες όχι βρισκόμαστε στην αρχή της συζήτησης ε, και πρέπει να προσέξουμε ώστε να έχουμε στην Ευρώπη ενιαία κατάρτιση των χρηστών. Έχουμε ενιαίους ελέγχους. Ε, θα το αμφισβητήσω αυτό. Ξέρω πόσο αυστηρή είναι η εκπαίδευση των γεωπόνων ε, στη Γερμανία για να επιτρέπεται να αγοράσει ένα τέτοιο προϊόν πρέπει να τεκμηριώνεται η αγορά. Ε, αμφιβάλλω αν αυτό γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι απομένουν πολλά να γίνουν στον τομέα αυτών. Όπως σας είπα, βρισκόμαστε στην αρχή της συζήτησης. Ε, δεν μπορούμε βιαστικά να λάβουμε απόφαση που να έχει ε, ευρείες συνέπειες ε, τις οποίες δεν θέλουμε. Ευχαριστώ, κύριος Κεπράντη. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Τζανόνι μίλησε για την έκθεση επικοινότητας που υιοθετήσαμε πέρυσι. και σύμφωνα με τη στρατηγική της Κομισιόν η ισολογική επικονίαση, η αξία της μάλλον, ορίζεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μεγάλο, μεγάλο ποσό. Άρα θα πρέπει να δοθεί αντίστοιχη αξία ενδιαφέρον. Ξέρετε, Πρόεδρε, πολύ συχνά με έχουν επικρίνει αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά επικρίνεται ότι αργεί, αργεί και καθυστερεί να λάβει αποφάσεις. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία εδώ να δείξουμε ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μπορεί να αντιδράσει γρήγορα. Είναι μια από τις περιπτώσεις ξεκάθαρες, οπότε μπορούμε να αντιδράσουμε έγκαιρα και γρήγορα και ίσως να είναι και αναγκαίο. Είναι κάπως περίπου χθε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος υιοθέτησε την έκθεση για ένα project που αφορά το πόσο α, δαπανηρό μπορεί να αποβεί η μη εφαρμογή της χρήσης ε, της προφύλαξης. Χαριστικό παράδειγμα εδώ. Δηλαδή, αν δεν δράσουμε τώρα σήμερα για αυτό το θέμα, μεθαύριο το κόστος μπορεί να είναι δυσβάσταχτο. Δύο ερωτήσει στην Κομισιόν. Σήμερα στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο ο αναπληρωτής υπουργό η αναπληρωτή υπουργό δήλωσε ή την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, στο Συμβούλιο Γεωργίας θα ζητήσει τη, τουλάχιστον την μείωση της χρήσης των νεονικοτιδών τη φιπρινόλη και ρωτώ, ξέρει κάτι παραπάνω ε, από εσάς ή είναι έτσι δική της πρωτοβουλία. Δεύτερο ερώτημα. Επίσης, έχετε καμιά εικόνα κατά πόσον έχει πιθανότητα να περάσει κάποια πρόταση από το Συμβούλιο. Και μάλιστα να πω κάτι ακόμη. Η Ολλανδή Υπουργό είπε ότι δεν υπάρχει συμφωνία στην Ευρώπη για μείωση τη χρήση αυτών των φυτοφαρμάκων, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η διαφορία, θα προβεί σε εθνικά μέτρα και ρωτώ νομικά είναι αυτό εφικτό. Ευχαριστώ. Και να ξαναδώσω το λόγο στην Εύσα και κατόπιν στον εκπρόσωπο από την Αυστρία εάν ε, θέλουν να απαντήσουν σε αυτά που ακούσανε. Nein. Εύσα, bitte. Η Εύσα, παρακαλώ. Um, I just wanted to point... Ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι στην Εύσα πραγματικά δουλεύουμε επί του θέματος το οποίο είναι πραγματικά πολυτομιακό. Γι' αυτό συστήσαμε μια task force, ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει όλες τις πτυχές του ζητήματος. Εντάχει θα ήθελα να απαντήσω ότι Πράγματι, εξετάσαμε όχι μόνο τις συνέπειες ε, στα, στον άνθρωπο, αλλά και τις συνέπειες στην ανάπτυξη των κοινοτήτων των ε, μελισσών. Όλα θα τα λαμβάνουμε υπόψη. Abschließend möchte der Kommission das Wort geben. Bitte, Herr Oui, merci, Monsieur le Président. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολλά τα ερωτήματα. Δεν ξέρω αν έχω αντίστοιχο χρόνο να απαντήσω. Έχουμε, πάρα, έχουμε όσο χρόνο θέλετε. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός χρονικός. Σας ευχαριστώ, Λίστα στα γερμανικά, εκπρόσωπος Κομισιόν. Λοιπόν, ένα ερώτημα το έθεσατε πολύ. Πρώτα απ' όλα ο κύριο Ντέιβις. Ποιο μέτρο είναι το κατάλληλο. Ποιο μέτρο θα πάρει η Κομισιόν. Α το πάρουμε από την αρχή το θέμα. Τέσσερις χώρες ήδη έχουν πάρει μέτρα. Δύο, το 2008, η Γερμανία και η Ιταλία. Και λάβουμε και εξηγήσει για τον Αραβόσιτο. Η Σλοβενία προέβη και αυτή σε μέτρα για όλους τους πόρους το 2008 και η Γαλλία πέρυσι το 2012 όχι για τον Αραβόσιτο Στη Γερμανία, μετά από περιπτώσεις ε, δηλητηρίασης ε, από μέλισσες, με την κανονική χρήση τέτοιων οικοτοδών. Είδαμε λοιπόν μαζική δηλητηρίαση ε, μελισσών. σε επίπεδο λοιπόν σχεδόν θανατηφόρο αυτή η δηλητηρία ε, χτύπησε τις ε, ε, κοινότητες των Μελισσών από τέσσερα διαφορετικά παραδείγματα. Οι Ολλανδοί φαίνεστε να είσαστε ανυπόμονοι από ό,τι κατάλαβα. Θα ζητήσετε να τεθεί στη μισή διάταξη ε, του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Δευτέρας από ό,τι κατάλαβα το θέμα αυτό. Και αν είναι αυτό η πρόταση της Υπουργού σα, γιατί δεν είναι πρόταση της Κομισιόν. Ακόμη η Κομισιόν δεν έχει συγκεκριμένη πρόταση. Οπότε είναι προφανές ότι κατα, κατανοώ ότι ο Ολλανδή Υπουργό απειλεί να πάρει εθνικά μέτρα. Ήδη άλλα τέσσερα κρατημέλη έχει πάρει εθνικά μέτρα. Εμείς δεν θέλαμε όμως να πάρουμε μέτρα κατά αυτών των τεσσάρων κρατών μελών. Ε, θεωρήσαμε ότι υπήρχε λόγος για τον οποίο πήραν αυτά τα τέσσερα κράτη-μέλη μέτρα ότι υπήρχε ε, τα στοιχεία από την επιστήμη ε, και η ΕΦΣΑ μας ε, έδωσε τα πρόσφατα πορίσματα της επιστημονικής κοινότητας, αλλά στις 16 Ιανουαρίου εμείς πήραμε μόλις τα στοιχεία της δηλαδή πριν από μια εβδομάδα. Η ΕΦΣΑ. Τη πήρε περίπου 9 μήνες λοιπόν της ΕΦΣΑ να απαντήσει στο ερώτημά μας. Δώστε μας και μας μία εβδομάδα τουλάχιστον, να προσπαθήσουμε να το σκεφτούμε ακόμα και αν δεν σκεφτόμαστε αρκετά γρήγορα. Εντάξει, δώστε μας ε, μια εβδομάδα, δέκα μέρες τουλάχιστον. Γιατί πολλοί από εσά ε, το είπατε, και ιδίω η κυρία Γκέρλινγκ, η απάντηση πρέπει να είναι αναλογική, ανάλογη μάλλον του προβλήματο. Η ΕΦΣΑ μας είπε ότι υπάρχουν φυτά που ελκύουν, προσελκύουν τις μέλισσες και άλλα όχι. Τα νεονικοτινοειδή ε, χρησιμοποιούνται και για τα, δύο είδη φυτών. Και για αυτά που ε, προσελκύουν ε, τις μέλισσες όπως το βαμβάκι, ο, ο, ε, ο ηλίανθος, αραβόσιτος, η ελαιοκράμβη. και με τον αραβόστο έχουμε και αυτή την έκκληση, την ακροή νερού από φυτό. αλλά υπάρχουν και άλλα φυτά που δεν προσελκύουν ε, τις μέλισσες όπως ε, είναι τα τέφτλα. Και εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε πώς ακριβώς ε, θα απαντήσουμε. Από την άλλη, σύμφωνα και με τις βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, ζητήσαμε από τις τρεις επιχειρήσεις, τις ενδιαφερόμενες, ε, μπάγερ και τα λοιπά, ζητήσαμε να δημοσιεύσουν ε, τις ε, παρατηρήσεις τους. Τους γράψαμε στις 16 Ιανουαρίου, την ημέρα δηλαδή που λάβαμε την γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ και τους δώσαμε διορία μέχρι τις 25, αύριο δηλαδή. Περιμένουμε λοιπόν την επίσημη απάντηση που θα έρθει να συμπληρώσει την συλλογική απάντηση της βιομηχανίας των ζανιοκτώνων που μας είπαν, όπως είπα και πριν, τα 50 εκατομμύρια ε, λοιπά. Θα έχουμε λοιπόν την μεμονωμένη απάντηση μία από αυτές τις τρεις επιχειρήσεις. για να εκφράσουν τη θέση τους απέναντι σε ένα τέτοιο μέρο που, μέτρο που θεωρείται σοβαρό. Η κυρία Κλάς μας ε, ζήτησε αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Είναι περίπλοκο το θέμα. Είδαμε ότι η Γερμανία και η Γαλλία απαγόρευσαν ε, την ε, επεξεργασία των ε, σπόρων αραβόσιτου και μόλις υπόθηκε ότι στην Ιταλία δεν υπήρξαν επιπτώσεις στην παραγωγή αραβόσιτου. Η Γαλλία το απαγόρευσε για την ελαιοκράμβη και μας είπαν ότι ούτε εκεί υπήρχαν σημαντικές επιπτώσεις, αλλά για την ελαιοκράμβη ένα τρίτο των, ε, των σπόρων ε, την χάνουν επεξεργασίες και τα δύο τρίτα όχι. Α, για τον αραβόστο. Επομένως, τώρα εξετάζουμε αυτό το ζήτημα της εναλλακτική ε, επεξεργασίας. Είναι δυνατόν, θεωρούμε. Θέλουμε μόνο να το παληθεύσουμε εάν μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί για τα φυτά που προσελκύουν τις μέλισσες, υπάρχουν εναλλακτικέ. Τώρα, για το ζήτημα της ε, σκόνης. Το εξήγησε και η ΕΦΣΑ, σας το ανέφερα και εγώ προηγουμένως. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να τη μειώσουμε αυτή τη σκόνη. Ε, στον, τη στιγμή της φύτευσης των κόκκων ή κάποιων άλλων σωματιδίων των συζανιοκτώνων, των νεονικοτινοειδών. Είναι σημαντικό και ε, σε αυτό το στάδιο λοιπόν να βρούμε μηχανήματα που να μπορούν να φυτεύσουν στο έδαφος ε, τους ε, σπόρους, τους επεξεργασμένους σπόρους, χωρίς να παράγουν ένα σύννεφο τοξικής σκόνης. Επομένω, σήμερα ε, δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω, εφόσον ακόμα το σκεφτόμαστε. Ακόμα και αν υπάρχει το θέμα αυτό με την Υπουργό ε, της Ολλανδίας, ούτε τη Δευτέρα λοιπόν δεν θα υπάρχει ζήτημα ε, ρύθμισης. Είναι πολύ νωρίς. Όμως θα δράσουμε σε δύο κατευθύνσεις. Ε, Πρώτον, έρευνα. Η ΕΦΣΑ και η Αυστριακή Οργάνωση ε, μας είπαν ότι υπάρχουν ε, κενά δεδομένων, data gaps, που πρέπει να συμπληρωθούν. Επομένως, ε, θα δούμε με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας πώς μπορούμε να αντετεκοποιήσουμε και να προωθήσουμε δύο προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή για τις μέλησες ή να εξετάσουμε νέα ε, σχέδια. Ε, μιλάμε για σχέδια που δεν είναι ιδιωτικά, γιατί υπάρχει και... Υπήρξε και αυτή η ένσταση αν πρόκειται για δεδομένα του, της φαρμακοβιομηχανίας ε, τα οποία δεν μπορούμε να πιστευτούμε πλήρως. Εδώ μιλάμε για έρευνες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη αλλά και από άλλους Φορεί, πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν ανεξάρτητα τα, τα στοιχεία και οι μελέτες. Ε, λογικά θα υπάρξει και μία νομοθετική δράση. Όμως δεν βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε θέση να σας πω κάτι. Δεν είναι επειδή θέλω να σας κρύψω κάτι. Απλώς δεν είμαι σε θέση να σας πω σήμερα ποια θα είναι τα σημεία που θα νομοθετήσουμε. Αυτή τη στιγμή τα σκεφτόμαστε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει, ε, δεν είναι κάτι επίγον. Ε, είναι χειμώνα, δεν βγαίνουν οι μέλισσε, μόνο κάνουν ε, μια βόλτα, αν θέλετε, όταν είναι ήπίε οι συνθήκες και επιστρέφουν κατευθείαν στην Κυψέλη. Αλλά δεν πρόκειται να, να πάνε στα άνθη αυτή τη στιγμή να επικοινωνιάσουν το ουσιαστικό αυτή τη στιγμή είναι η... θα ξεκινήσουν οι καλλιέργειες αραβοσίτου τον Μάρτιο-Απρίλιο, ανάλογα με την ε, περιοχή. Και δίκα σε αυτές τις καλλιέργειες αραβοσίτου έχουν ήδη ε, προετοιμαστεί ε, οι κόκκι αυτοί οι σπόροι. Γιατί το 1 τρίτο αυτών των σπόρων, των κόκκων, έχουν καλυφθεί έχουν μια επικάλυψη οικοτεδιδών. Έχει γίνει ήδη αυτή η προετοιμασία. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια εκτίμηση του προβλήματος. Έχουμε ας πούμε κάποιες εβδομάδες για να ολοκληρώσουμε αυτή την νομοθεσία, να διαβολευτούμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους γεωργούς βεβαίως. Είναι οι πρώτοι και άμεσα ενδιαφερόμενοι. Με τη βιομηχανία των Συζανιοκτώνων με τους μελισσοκόμους και με τους Γιωργούς γιατί και αυτοί εμέσως επηρεάζονται, και με τις αρχές των κρατομελών και τις πολιτικές αρχές. Έχουμε λοιπόν κάποια ζητήματα να διευθετήσουμε. για να είναι όλα ξεκάθαρα, ας πούμε τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως ε, θα εξακολουθούμε να αναλύουμε ε, τις επιπτώσεις, να, δούμε πώς, να βλέπουμε πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις ε, δράσεις μας, γιατί δεν θέλουμε να, η απάντηση μας να είναι και δυσανάλογη. Η ΕΨΑ μας είπε ότι υπάρχουν πέντε νέων νοικοτονοειδή. Υπάρχουν δύο ακόμα τα οποία δεν έχουμε μελετήσει ακόμα, αλλά φαίνεται ότι είναι λιγότερο προβληματικά. Αλλά καλό θα ήταν να θέσουμε το ερώτημα στην ΕΦΣΑ για να διευκρινιστεί και αυτή η κατάσταση. Υπάρχει μια έκτη ουσία που δεν είναι νέο νοικοτινοειδή, το φιπρονίλ, για την οποία ζητήσαμε αξιολόγηση από την ΕΦΣΑ, η οποία όμως θα μας έρθει λογικά τον Μάρτιο του 2013. Αν είναι αρνητική η, η εκτίμηση αυτή, η αξιολόγηση, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να πάρουμε μέτρα για το φιπρονίλ. Θα περιμένουμε όμως τη γνωμοδότηση της ΕΡΣΑ το Μάρτιο. Η κυρία Κλάς ε, ανέφερε ένα σημαντικό θέμα, ότι δηλαδή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι μέλισσες κατά την αξιολόγηση του κινδύνου, την εκτίμηση του κινδύνου των ζυζανιοκτώνων. Πράγματι αυτό είναι θεμελιώδους σημασία και ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ, γιατί Πράγματι, αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν και σιγά σιγά αναπτύχθηκε αυτή η ιδέα. Ζητήσαμε λοιπόν από την ΕΦΣΑ να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τον κίνδυνο, ειδικά για τις μέλισσες και όχι γενικά για το περιβάλλον και για το περιβάλλον γενικά βέβαια, αλλά πιο συγκεκριμένα και για τις ε, μέλισσες. Η ΕΦΣΑ λοιπόν θα μας δώσει ένα έγγραφο για τους ε, ειδικού κινδύνους ε, των ζανιοκτώνων για τις μέλισσες τον Μάρτιο, το Μάιο, ε, για το 2011 τα υπόθηκαν πράγματι το πρόβλημα του συνδρόμου της ε, κατάρρευσης των των απικιών είναι πράγματι απαρτίζεται από πολλούς παράγοντες. Ε, ε, περιβαλλοντικοί παράγοντες, ασθένειες, ε, αγροτικές πρακτικές, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Πρέπει να αξιολογήσουμε λοιπόν το σύνολο αυτών των παραγόντων. Όμως, αυτή τη στιγμή ε, τα ζανιοκτώνα και συγκεκριμένα τα νεονικοτινοειδή θεωρήθηκαν σημαντικός παράγοντας αυτής της ε, σχεδόν θανατηφόρας τοξικότητας, είναι κάτι που βεβαίως και εξετάζουμε, όπως ε, οι ασθένειες. Διάφορες ασθένειες που μπορούν να έχουν οι μέλισσες, είναι σημαντικό βεβαίως να τις καταπολεμήσουμε με το πρόβλημα της ε, μη διάθεσης ε, συγκεκριμένων φαρμάκων. Ήταν δύσκολα αυτά τα ζητήματα. Ακόμα πιο περίπλοκες είναι οι γεωργικές πρακτικές. Όμως αυτή η στρατηγική για την υγεία ε, των μελισσών που παρουσιάσαμε με τους συναδέλφους μαζί και με τις άλλες γενικές διευθύνσεις ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό κείμενο όπως ανέφερε η κυρία Βελή. point euh, de M. sur... Τώρα ένα σημείο του κυρίου Χρυσόγελου για, τα, ε, για, για τις επιπτώσεις της ε, επεξεργασίας ε, για ένα άλλο έντομο που εντοπίζεται στους Φινικές και καταστρέφει τους φοίνικες που βρίσκονται και απαντώνται σε όλες Τη ε, πόλη σε όλα τα τοπία της Μεσογείου. Είναι λοιπόν ένας μεγάλος σκαραβαίο ε, που καταστρέφει τους φίνικες. Πράγματι, αν ε, εδώ πέρα χρησιμοποιήσουμε ζυζανιοκτώνα, όταν υπάρχουν άνθη που προσελκύουν τις μέλισσες για να σκοτώσουμε αυτό το σκαραβαίο, δεν θα σκοτώσουμε το σκαραβαίο, σκοτώνουμε και τι μέλισσες. Ούτε αυτό είναι καλό. Υπάρχουν λοιπόν κάποιε πρακτικές, δηλαδή να κόψουμε δηλαδή, τα άνθη των ε, φινίκων, γιατί στην ε, Μεσογειακή Ευρώπη... Πώς θα... Δεν υπάρχουν ε, οι καρποί, ε, οι χουρμάδες είναι ε, κάτω στις ε, βόρειες ακτές της Αφρικής. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να κόψουμε τα άνθη για να προστατεύσουμε ε, και το δέντρο και τις μέλισσες. Είναι λοιπόν δυνατόν να ακολουθήσουμε αυτή την πρακτική. Bon, Monsieur Poch nous a dit que nous avons changé d'avis. Είπατε ότι θα αλλάξουμε άποψη, θα αλλάξουμε γνώμη. Είναι πράγματι, συνάδελφε, γιατί οι δύο οργανισμοί μας έδωσαν επιστημονικά στοιχεία. Είναι δύσκολο για την Επιτροπή να ενεργήσει βάσει εντυπώσεων ή συναισθημάτων ή εκθέσεων των μελισσοκόμων. Πράγματι, οι μελισσοκόμοι εδώ και δέκα χρόνια περίπου είχαν εντοπίσει τον κίνδυνο των νεονικοτινοειδών. Στη Γαλλία, θυμόμαστε ότι υπήρχαν ε, ε, διαμαρτυρίες εδώ και πολλά χρόνια για αυτές τις ουσίες, αλλά χρειαζόμασταν αποδείξει και δεν ήταν εύκολο να τις συλλέξουμε. Χάρη σε αυτές τις τρεις ε, μελέτες, τη γαλλική, τη βρετανική και τη γερμανική, στις αρχέ 2012, ε, συλλέξαμε εν μέρη τονίζω αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία γιατί και η ίδια η ΕΦΣΑ λέει ότι υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και αλλάξαμε γνώμη ακόμα και αν μπορούσαμε να υποπτευθούμε ε, ε, τις αρνητικές επιπτώσεις των νεονικοτενοειδών, ε, πρέπει πάντα να βάλουμε υπόψη και τον βαρύ αντίκτυπο ε, αυτών των μέτρων για τους γεωργούς και για τη βιομηχανία και δεν μπορούμε να τα στηρίζουμε όλα αυτά σε εντυπώσεις. Πρέπει να υπάρχουν ε, αυτές ε, επιστημονικές αποδείξεις για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την αρχή αυτή ε, της πρόληψης. Και ε, θα μας πει, ακόμα και η μηχανία μας λέει ότι ε, ναι, η ΕΦΣΑ δεν σας έχει δώσει αρκετά στοιχεία, μην κάνετε τίποτα. Όμως εμείς, εν μέρη τουλάχιστον, θα αξιοποιήσουμε αυτή την αρχή. την αρχή της προφύλαξης λοιπόν. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε, απαντώντας ε, προς, τους, ε, προς τα μέλη της Επιτροπής σας. Αν όμως έχω ξεχάσει κάτι, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ja, wünscht der Fragesteller noch das Wort? Chris Davis, bitte. Ο Chris Davis θέλει το λόγο, παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Ναι, καταλαβαίνω το νόημα αυτών που λέει η Επιτροπή, αλλά όλο λέτε, σκέφτεστε, αξιολογείτε, θέλετε περισσότερες έρευνε, περιμένετε την ΕΦΣΑ, αλλά απ' την άλλη πρέπει ταυτόχρονα να ενεργήσετε άμεσα. Δεν έχω καταλάβει πότε θα γνωρίζουμε αν θα εισάγετε νομοθετικέ προτάσεις. Écoutez les conclusions du Conseil d'Agriculture de Να περιμένετε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Δευτέρας.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 Μια σύντομη αναφορά. Ακούσαμε πολλά από την Κομισιόν και από την ΕΦΣΑ. Η Κομισιόν μας είπε ότι μέχρι το 2012 όλα ήταν ανθυρά και ρόδινα. Να λέγω από το 2003 έχω στοιχεία που υπήρχαν προβλήματα. Ήδη το 2003 επιστημονικά ιδρύματα, μιλάμε για ιδρύματα των ΙΠΑ, και, και εσείς είπα υπάρχει επιστήμη, έτσι, λοιπόν, και ξέρετε τι λέει ότι αυτή η ουσία είναι ιδιαίτερα τοξική για τις μέλισσες και υπάρχει το δυναμικό χρόνιας και οξίας ε, ε, δηλητηρίασης μελισσών καθώς μεταφέρονται υπολείμματα ε, στο μέλι και στο νέκταρα των μελισσών και αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε σχεδόν θανατηφόρα συμπτώματα και επηρεάζει δραστικά την αναπαραγωγική δυνατότητα των μελισσών. Όχι λοιπόν ότι τώρα εμφανίστηκε το πρόβλημα το 2012 και όλα ήταν καλά έω τώρα και οι επιστήμονε μας είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολύ νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο? Όχι. Να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν στη συζήτηση και τον κύριο Πουλέη και την ομάδα του Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Ντέιβις. Ε, πάντω είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προφορική αυτή ερώτηση και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι σημερινε προκλήσεις και ευκαιρίες για την ενέργεια από ανανεώσιμες ε, πηγές στην Ευρωπαϊκή Αγορά ενέργεια. Ε, η κυρία Κούκοβιτς δεν μπορεί να είναι παρούσα, γι' αυτό προτείνω να συζητήσουμε το θέμα κάποια άλλη στιγμή. Ε, θα έχουμε και την ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 29 Ιανουαρίου και η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, στις 19 Φεβρουαρίου θα ψηφίσει. Ε, η, στην Ήτρε θα ψηφίσει 18 Μαρτίου και από ό,τι φαίνεται ε, η έκθεση θα μπει στην Ολομέλεια του Απριλίου. Oh. Yeah. Η 29, das 29 είναι η δική μου έκθεση, σχεδόν την ξέχασα ε, και έχει να κάνει με την ε, οδηγία του πρωινού τη λεγόμενη. Έχει να κάνει με τα προϊόντα του πρωινού, ε, καφέ, κακάο, σοκολάτα, ε, μέλια, γάλα καθώς ε, και το ε, γάλα. Δεδομένης της ε, συνθήκης της Λισαβόνας είναι απαραίτητο να γίνει μια προσαρμογή ε, που έχει να κάνει με τις κατεξουσιοδότηση νομικές πράξεις. Ε, σύμφωνα με το άρθρο 290. Ε, ε, χωριστή και κατά την εξέταση ε, κατάλαβα ότι δίνουμε σημαντικές εξουσίες στην Επιτροπή όσον αφορά την περιγραφή των προϊόντων αυτών, ε, αν ακολουθήσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και στην ε, οδηγία για τους ε, χυμούς των φρούτων ε, συνεννοηθήκαμε συμφωνήσαμε πώς ε, θα προχωρήσουμε και ε, ως ε, εισηγητής παρακολούθησα τη ε, διαδικασία της έκθεσης αυτής και στις 28 Νοεμβρίου βρήκαμε είδαμε ευρία υποστήριξη από τους συναδέρφους για την οδηγία αυτή. Το Συμβούλιο συζητάει αυτή τη στιγμή επίσης το σχέδιο και φαίνεται να ακολουθεί τη δική μας γραμμή ώστε οι κατεξοδότηση πράξεις να περιοριστούν σε κάποια μη ε, ουσιαστικά στοιχεία. Θα ήθελα πριν την Ολομέλεια να προσπαθήσω μαζί με τους κοιόδης εισηγητές ε, να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό θα πρέπει να είναι δυνατόν, διότι ουσιαστικά δεν υπάρχει διάσταση απόψεων. Και περιμένω εναγωνίως ε, να ακούσω τη συζήτηση. Η κυρία Κλάς εκπροσωπεί την κυρία Οκονή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Η Σοφία Οκονή ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρούσα. Και αυτή τονίζει ότι είναι σημαντική η έκθεση αυτή. Ε, και με τις κατεξουσιοδότηση πράξης ε, έχουμε τώρα ένα μόνιμο καθήκον να ορίζουμε πώς θα εφαρμόζεται και θέλουμε να τονίσουμε ότι στην ε, οδηγία αυτή όταν μιλάμε για ουσιαστικές ε, τροποποιήσεις στη βασική πράξη τότε αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο τέτοιες μεταχείριση. Η κυρία Οκονή συμφωνεί με τον εισηγητή Πιστεύει ότι είναι καλές οι τροπολογίες και τη Σερενάτε Σόμερ και του Ζαν Πιεροντή. Η Σοφή βλέπει κάπως επιφυλακτικά την τροπολογία της Λίντα Μακέβαν. καθώς και την τροπολογία Ούτσκι στις τροπολογίες 20 και 21 Η Λίντα Μακέβαν θέλει να μπορεί να γίνει προσθήκη, όχι όμως σε διαγραφή ε, των ε, στοιχείων στο παράρτημα. Ε, αυτό δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά. Γιατί δηλαδή να μπορεί κανείς να κάνει το ένα και όχι το άλλο. Πάντως γενικά η Σοφία Κονή στηρίζει τη γραμμή του εισηγητή και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να γίνει αυτή η συνάντηση που λέτε με τους κοιόδες εισηγητές. Ε, ευχαριστώ κυρία Ράιμερς. Ε, ναι, δεν ε, μου απομένει τίποτα άλλο από το να συμφωνήσω. Στηρίζουμε τη γραμμή του εισηγητή και προσβλέπουμε στην ε, συζήτηση περί συμβιβασμού. Πιστεύω ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Αχ, τέτοιες, παρεμβάσεις θα ευχόμουν να είχα και νωρίτερα. Ο Μπαρτ ε, Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Σας στηρίζουμε πλήρως ως ε, εισηγητή. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. So, dann, äh, ε, habe ich Frau Liotard? Da haben wir sonst noch Wortmeldung. Nein, da möchte der Kommission. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Να ακούσω τι θα μου πει, μάλλον θα της αρέσει η γραμμή μας. Nee, ah, nee. Sachstand. Ah, das ist ein Sachstandsbericht. Ja. Uh, Πρόεδρε, χαιρετίζουμε την έκθεση. Και δεν θέλω τώρα να σας χαλάσω και το πάρτι για αυτή την ευρεία συμφωνία. Όπως είπαμε και την άλλη φορά, η Κομισιόν παραμένει πεπισμένη ότι χρειάζεται πράξη κατεξιοδότηση για να μπορεί να, προσαρμόζει τεχνικά και μη ουσιώδη στοιχεία της πρότασης και να μπορεί να αντιδρά γρήγορα, κατάλληλα και κατά κύριο λόγο αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά το κόστος. Διότι όταν ακολουθούμε την ε, κανονική διαδικασία για να προσαρμόσουμε τεχνικές λεπτομέρειες, αυτό είναι κάτι χρονοβόρο ε, και δαπανηρό. Υπ' αυτή την έννοια λυπούμεθα λοιπόν, ιδιαιτέρως, γιατί το σχέδιο έκθεσης του Κοινοβουλίου καταργεί και κείμενα σε της κομισιών αναφέρουμε στην Οδηγία 2036 παράρτημα Β σχετικά με τα το συστατικά του κακάου και σοκολάτας. Μιλάμε επίσης ε, για τον κανονισμό 114-2000 ε, για το αφιδετωμένο γάλα και εκεί μας έχουμε άλλες εξουσίες που τις ακυρώνονται σήμερα. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για την μαρμελάδα, 113 του 2001 και εσείς θέλετε να κρατήσετε το παράρτημα 2 γιατί τα συστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επί πρόσθεσης μαρμελάτα στη βασική πράξη για τους χυμούς φρούτων. Ενώ πρόσφατα και η οδηγία και έχει ε, κατά πράξη καταξιοδότηση εξουσίας αντίθεση με αυτό που λέτε εσείς στην εκθέση. Υπ' αυτή Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό που λέτε, εμείς χαιρετίζουμε την τροπολογία 20 Τη κυρία Μακέβιν, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα σωστή κατεύθυνση, η οποία πολύ ορθά λέει ότι σε περίπτωση αλλαγών συνταγών για τη μαρμελάδα, μια γρήγορη τροποποίηση του ε, ε, ανοιχτού καταλόγου είναι κάτι επιθυμητό. Και αυτό δεν είναι δυνατόν με την ε, τακτική νομοθετική διαδικασία. Σας παρακαλώ να θυμάστε ότι η πλαίσια επιτρέπει στον νομοθέτη να επιτρέψει στην Κομισιόν να τροποποιεί τεχνικά μειωσιώδη στοιχεία όπως είναι διάφορα ποσοστά επιξηρού ή πυγρού, ο βαθμός φουλαρισμού στα, στα, στη ζάχαρη κτλ. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό προτείνεται υπερβολικά χρονοβόρο και δαπανηρό αν πρέπει να ακολουθούμε πάντοτε την τακτική νομοθετική διαδικασία για αυτά. Τώρα για τα δικαστικά ζητήματα και για την προτινόμενη περίοδο πενταετίας πράξη καταξιοδότηση, με την υποβολή εκθέσεων που μας καλείται να κάνουμε, εμείς θεωρούμε ότι σε ό,τι αφορά αυτές τις οδηγίες, τα χρονικά όρια και η υποβολή εκθέσεων θεωρούμε ότι είναι κάτι μη αναλογικό βάσει προτεραιότητα εμπειρίας καθώς πολύ λίγες ήταν που έγιναν μέσα στον χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, δεν είχαμε τελείως αρμονική ατμόσφαιρα σήμερα. 19 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια του Απριλίου μάλλον θα έχουμε το θέμα στη μέση διάταξη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις αυτές. Περνάμε στο επόμενο θέμα της μέσης διάταξης. Ε, το επόμενο θέμα είναι το υπαριθμό 31. Κατάσταση προόδου όσον αφορά τη δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα, CCS. Να δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον Chris Davis, που είναι εισηγητή. Παρακαλώ. Thank you, Chairman. Uh, delighted that Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ακόμη έχουν παραμείνει αρκετοί συνάδελφοι για αυτό το τόσο δύσκολο θέμα τέτοια καθυστερημένη ώρα. Έως το 25% των παγκόσμιων εκπομπών και όλες τις εκπομπές από τη βιομηχανία, χημική βιομηχανία, χάλιβα κτλ. Αλλά χωρίς να δίνουν πραγματικές εναλλακτικές. Είναι πραγματικά λυπηρό. Γίνεται πάρα πολλή δουλειά προσπάθεια να αναπτύξει τεχνολογία ε, στον κόσμο, αλλά γίνεται προσπάθεια και στην Ευρώπη και στην Κομισιόν. Ε, και κοιτώ και την εκπρόσωπο του ΔΕΛΤΑ Ενέργεια και Κλίματος, που προσπαθούν να προωθήσουν τα project CCS. Αλλά τα αποτελέσματα είναι πολύ απογοητευτικά. Πρόσφατα είχαμε την ανακοίνωση για το ε, μηχανισμό κατανομής 300. Σας παραπέμπω σε αυτό που είχαμε πει το 2008 και καταφέραμε να πείσουμε το Συμβούλιο να δεχτεί αυτή την έννοια. Αυτός ο μηχανισμός είχε σκοπό να δημιουργήσει συνολικά 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δύο τρίτα εξ αυτών ε, των πιστώσεων οδήγησαν σε 1,5 δις. Και αρχικά κρατημέλη ήθελαν αυτά τα χρήματα και τελικά που καταλήξαμε πριν τα Χριστούγεννα. Να προωθηθεί ένα ακόμη μονομένο project CCS. Κανένα πρόβλημα με τα χρήματα που πάνε σε ένα καινοτόμο project, αλλά το βασικό μας πρόβλημα ήταν ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου η νέα τεχνολογία. Και αυτό οδήγησε σε ένα μεταξύ αυτών και η τιμή του άνθρακα που συζητούσαμε και το πρωί. Αυτές οι πιστώσει ε, οι 300 πιστώσεις δεν είναι τίποτα ουσιαστικό, τίποτα σημαντικό ως μηχανισμό χρηματοδότησης. Τα διαθέσιμα ε, χρήματα ε, και τα έσοδα από τις, από τις τελικά δεν είναι αυτό που περίμεναν τα κράτη-μέλη. Οπότε το κόστος της στάθμισης δεν ήταν τελικά αυτό που προσδοκούσε κανεί. Μεγάλη απογοήτευση και ρωτούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Το Μάρτιο 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι θέλει τουλάχιστον 12 project CCS έως το 2015. Και ένα να εγκρίνουμε, τυχεροί θα είμαστε έως τότε. Οπότε κοιτάξτε τριγύρω και σκεφτείτε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε δύο γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν, δύο προσώπους εδώ και το πρώτο ζήτημα είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα για αυτή τη δεύτερη φάση των 300 πιστώσεων. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ελπίζαμε να μπορέσουμε ε, να φτάσουμε και τις 900.000 ευρώ ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε 300 εκατομμύρια ευρώ για ε, συγχρηματοδότηση. Πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Λίγε χώρε έχουν μείνει και η Ιταλία δεν φαίνεται να μπορεί να προωθήσει το project τη. Η Γερμανία ούτε καν ενσωμάτωσε την νομοθεσία του 2008-2009. Το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται ότι είναι ανίκανο να ανταποκριθεί στο ευρωπαϊκό χρονοδιάγραμμα, ακόμα και αν αξίζει τη χρηματοδότηση. Φαίνεται ότι μόνο μόνο η Ολλανδική κυβέρνηση θα προχωρήσει. Αλλά αυτή η κατάρρευση της τιμής του άνθρακα σήμερα που έφτασε στα 2,6 ευρώ στον τόνο, τι σημαίνει, ότι ουσιαστικά είναι άνευ αξίας αυτό το, αυτό το ταμείο. Οπότε και η όλη ανακοίνωση της έναρξης διαδικασίας δεν έχει νόημα, γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα καταλάβει ότι τελικά μιλάμε για ένα σημαντικό project το οποίο δεν μπορεί όμως να ξεκινήσει τώρα λόγω των τιμών. Η ΓΑΜΑ ΔΕΤΑ Ενέργειας προετοιμάζει μία ανακοίνωση για να προωθήσει το CCS. Έχουμε δει ανεπισήμως κάποια σχέδια αυτού του κειμένου. Ακούγονται κάποιες ιδέες για μια ρυθμιστική προσέγγιση. Εγώ να ακούσω από την Κομισιόν να μας πει πότε θα το έχουμε αυτό το κείμενο να το συζητήσουμε. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν και άλλες ιδέες. Για παράδειγμα, ιδίω οι συμπράξει μεταξύ κυβερνήσεων, γιατί ένα project CCS κοστίζει πάρα πολλά, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούν οι κυβερνήσεις, άρα να δώσουμε κίνητρα στις κυβερνήσεις για να υπάρξει συνεργασία. Αυτά, να σταματήσω εδώ. Απλά να πω ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η τεχνολογία δεν βλέπω να υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε από την αθρέα προσέλευση εδώ. Όλοι μιλάνε για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ε? για ολική ενέργεια κτλ. Τα διάφορα λόγια αυτά πιέζουν. Αυτή η τεχνολογία όμω είναι πολύ σημαντική γιατί αν θέλουμε να έχουμε μόνο των ε, εργοστασίων και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα ορυκτά καύσιμα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ακούσω την Κομισιόν. Kollegin Συνάδελφο Καρτίνη, συνάδελφε Τέιβις, μόνο εσείς έχετε απομείνει μου φαίνεται. Κυρία Καρτίνη, σας ρωτώ προσωπικά, θέλετε το λόγο. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Αλλιώς θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Όχι. Απλά να πω ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον Κρις Davis. Σε κάποιες φορές δεν ταυτίζονται οι απόψεις μας. Ας πούμε στο ETS δεν ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Είναι προφανές όμως ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι μείζωνο σημασία. χωρί τεχνολογία ε, CCS, πολλοί από τους στόχου που έχουμε θέσει δεν ε, μπορούμε ούτε καν στο όνειρό μα να τους επιτύχουμε στην Ιταλία. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό project που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, αντιμετωπίσαμε σημαντικά προβλήματα Όσοι έχουν ευαισθησία για το περιβάλλον, συχνά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν στη τεχνολογία CCS ότι είναι το κατάλληλο εργαλείο για να επιτευχθούν οι στόχοι που θέλουμε λόγω της οικολογικής ευαισθησίας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που θέτουν το πρόβλημα, άτομα που είναι πολύ δραστηριοποιημένα, για την προστασία του περιβάλλοντος και για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι, μετά είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ε, μπαίνουν πίσω από δοφράγματα για να μην χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες όπως τεχνολογίες SES. Υπάρχει η αίσθηση ότι αυτή η τεχνολογία αντίκειται στις ε, περιβαλλοντικές πολιτικές. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό να σκεφτούμε και μία εκστρατεία ενημέρωσης, μια ξεκάθαρης μια κάθαρης ηχηρής ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη για αυτό το ζήτημα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ουσιαστικά είμαστε ενώπιον ενός παραδόξου. Ευχαριστώ πολύ. Στην πατρίδα μου δυσκολευόμαστε με τα θέματα του CCS, ιδιαίτερα της αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά βέβαια όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και με το θέμα που συζήτησαμε σήμερα το πρωί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλή η ιδέα να ε, χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα αυτά. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να έχουμε το CCS σε εργοστάσια παραγωγή ρεύματο, αλλά σε άλλου τομεί, όπω είναι η παραγωγή ατσαλιού και άλλου τομεί, ε, χρειαζόμαστε ε, κάτι τέτοιο. Βρίσκω ότι είναι ε, λυπηρό το ότι έχουμε φτάσει στην κατάσταση αυτή, το ότι ε, πραγματοποιήθηκα ένα πρόγραμμα ενώ στόχος ήταν κάτι άλλο. Αλλά το, το CCS, η αποθήκευση και η, η δέσμευση και αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα συνδέεται και με την τιμή του διοξιδίου του άνθρακα. Ε, ήθελα σχεδόν να ρωτήσω του αδέρφου αν θέλει κανεί άλλο το λόγο, αλλά έχουμε μόνο δύο εδώ πέρα. Να δώσω το λόγο στην Κομισιόν τον κύριο Τουλιέ, που είναι επικεφαλή. Ε, της ε, μονάδας ε, και διευθυντή για τι ε, ε, ε, χαμηλού άνθρακα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Σα ευχαριστώ που προσκαλέσατε την Επιτροπή σε αυτή τη συζήτηση για το CCS. Υπάρχουν πολλά ζητήματα σχετικά με την τεχνολογία και το μελλοντικό τους ρόλο στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει ούτε ένα project τέτοιο στην Ευρώπη. Παρόλα όσα είχαμε ακούσει για πολλά project το 2015, ήδη αναλύουμε τους λόγους για τους οποίους η τεχνολογία CCS δεν έλαβε τη βράβευση υπό το ε, πρόγραμμα της χρηματοδότηση αυτό το 300. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά, σημαντικά χρηματοδοτικά μέσα ε, που θα μπορούσε να πάρει ένα σχέδιο από την πιλωτική του φάση προς την ε, εμπορική ανάπτυξή του. Και βρισκόμαστε στο στάδιο που οι πληροφορίες για, τη, για τις πρώτες προτάσεις για το 9300 συζητούνται. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2012 και είναι αλήθεια ότι από, τα, τις δύο τεχνολογικές ομάδες, το CCS και ε, τα καινοτόμα ανανεώσιμα, ε, το δεύτερο μόνο έλαβε το βραβείο του 1,2 δις ευρώ. Η προκατακτική ανάλυση των ε, υποψηφίων, και είναι σημαντικό και αυτό να το έχουμε κατά νου, δηλαδή ποιο ήταν το ενδιαφέρον που εκφράστηκε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του προγράμματος 2010, ήθελα να σας πω ότι λάβαμε 13 αιτήσει για τις χρηματοδότηση των προγραμμάτων CCS. Ήταν σχεδόν ο στόχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 13 projects σε όλες τις κατηγορίες της τεχνολογίας και ήταν ε, πολύ θετικό που είδαμε ότι ήταν πολύ καλής ποιότητας ε, αυτές οι προτάσεις και τεχνολογικής οριμότητας και στηρίζονταν από τα κράτη-μέλη. Τώρα μιλάμε για το 2010. Ολόκληρη διαδικασία της ε, αξιολόγησης αυτών των προγραμμάτων μας πήρε δύο χρόνια και πέρασαν όλοι. Επομένω, όλα έβαιναν καλώς με αυτά τα προγράμματα. Όμως η διαδικασία υπό το πρόγραμμα απαιτούσε μια τελική επιβεβαίωση από τα κράτη-μέλη που υποβάλλουν τις αιτήσει για συγχρηματοδότηση. Και εκεί απέτυχαν αυτά τα project. Όλα εκτός ε, από ένα δεν επιβεβαιώθηκαν. Ένα μόνο επιβεβαιώθηκε από το κράτος μέλος και στη συνέχεια επεσήρθη μετά από μερικές εβδομάδες αρχίσαμε να κάνουμε ερωτήσεις και να αναλύουμε τους ε, λόγους, τις αιτίες για αυτή την έλλειψη τελικής επιβεβαίωσης. Και σήμερα, αυτό που μας είπαν και τα μελη μπορούμε να σας πούμε λοιπόν, ότι η αιτία μια επιβεβαίωση στο project του τελευταίο στάδιο ήταν ότι δεν υπήρχε εθνική χρηματοδότηση ή φορείς Υπήρχαν καθυστερήσεις και στις διαδικασίες αδειοδότησης ε, σε κάποια κρατημέλη γιατί είναι περίπλοκα αυτά τα project ε, και απαιτούν ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών αδειών οι οποίες καθυστέρησαν σε ορισμένες περιπτώσεις ή δεν δόθηκαν καθόλου. Υπήρξε και περίπτωση συνεχιζόμενου εθνικού διαγωνισμού που έτρεχε παράλληλα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αλλά δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως για να μπορέσει το κρατός μέλος να επιβεβαιώσει ένα-δύο παραπάνω project. Και τέλος, άλλος λόγος θα μπορούσε να είναι ε, οι προβλέψεις για την τιμή του άνθρακα, αλλά δεν ήταν λόγος αυτός να μην επιβεβαιωθούν τα προγράμματα. Η Επιτροπή προετοιμάζει έκθεση για την ε, Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής, όπου αναλύονται ενδελεχώς ε, οι αιτίες αποτυχίας αυτού του προγράμματος και πράγματι πάντα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει λοιπόν μια δεύτερη πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του προγράμματος 9300. Δεν έχει τεθεί ακόμα ημερομηνία έναρξης αυτής της πρόσκλησης. Πρέπει να γίνουν ακόμα κάποια απαραίτητα βήματα προς τα εκεί. Έχουμε πρώτα απ' όλα την ε, συνάντηση αυτή την κλιματική αλλαγή και τη συζήτηση με τα, κράτη, μελη Είναι δύσκολο λοιπόν ε, να πούμε σήμερα πότε ακριβώς θα γίνει αυτή η πρόσκληση. Βεβαίω πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη πρόσκληση παρά τις υψηλές προσδοκίες ε, για το ποσό, από τα 4 εκατομμύρια δηλαδή που αναμέναμε αρχικά φτάσαμε στο 1,5, Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι η πρώτη πρόσκληση ήταν ε, επιτυχής γιατί Πράγματι, ορισμένα project έχουν τύχει σε χρηματοδότηση και από τα 27 κρατημέλη, τα 16 βρίσκονταν στην ομάδα των κρατών που ε, έλαβαν αυτή τη βράβευση από το NER 300. Αυτά από τη μία πλευρά. Από την πλευρά πολιτική τώρα, ε, προετοιμάζουμε έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας ε, CCS που προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και αναμένεται φέτος αυτή η έκθεση. Θα είναι μια καλή δυνατότητα να εξετάσουμε σε βάθος ε, τους ε, λόγους πολιτικής ή εφαρμογής ε, που εξηγούν γιατί δεν έχει φτάσει στο εμπορικό επίπεδο η εφαρμογή του CCS. Πρέπει να έχουμε κατά νου αναλύσεις της πρώτης φάσης του προγράμματος του NER 300 και η σε βάθος ανάλυση της εφαρμογής ε, της οδηγίας θα μας δώσουν μια ξεκαθαρή εικόνα για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ε, στο άμεσο μέλλον για να γίνει απόλυτα εμπορική και λειτουργική ε, αυτή η προσέγγιση του CCS. Να δώσω τώρα τον λόγο στον συνάδελφο Hans von Stein για σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και τον Hans Mansfield από την ε, Κομισιόν, ε, από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω μόνο τον συναδελφό σχετικά με την ε, υποστήριξη αυτού του project. Προβλέπετε μία ανακοίνωση από πλευράς μας. Πρότεινε λιγανάστε για το CCS στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ανακοίνωση που ήδη περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα εργασία της Κομισιόν για το 2012. Τελικά όμω αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερα να περιμένουμε. Να δούμε πρώτα απ' όλα τα αποτελέσματα τη πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντο και μετά να προβούμε στην ανακοίνωση. Τώρα που είδαμε τα αποτελέσματα και εμείς συμμεριζόμαστε την ίδια απογοήτευση με τον Chris Davis σε ό,τι αφορά το CCS αυτού του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανησυχίες έχουμε και για τα project που επελέγησαν με βάση το οικονομικό πρόγραμμα για ανάκαμψη. Αρχικά έξι CCS project CCS μεγάλης κλίμακας. Το ένα επισήμως έκλεισε, σταμάτησε, το γερμανικό. Και τα άλλα πέντε projects, όπως είπε και ο κύριος Davis, έχουν πολλά ερωτηματικά. Σοβαρές λοιπόν ανησυχίε. για το CCS στην Ευρώπη Γι' αυτό δουλεύουμε αυτή την ε, ανακοίνωση ακόμη. Ξέρω ότι κάποιοι έχουν διαρρεύσει διάφορες εκδοχές του κειμένου. Λοιπόν, εγώ το μόνο που επιβεβαιώνω είναι ότι δουλεύουμε πολύ σκληρά για να τελειώσει η σύνταξη της ανακοίνωσης το μότερο δυνατόν. Είναι πολύ σημαντική η ανακοίνωση κατά τη γνώμη μας, ιδίως λόγω της παρούσας κατάστασης φαίνεται τουλάχιστον πρόθεσμα να υπάρχει μια στροφή στα ορυκτά καύσιμα τουλάχιστον για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Παρότι έχουμε τόσες εξελίξεις με το σχεδοστολιθικό, άντακα και άλλα πράγματα αλλού στον κόσμο στη ΣΥΠΑ. Ίσως λοιπόν τελικά οι εκπομπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξηθούν. λόγω του ότι είναι, θα είναι μεγαλύτερο το μερίδιο της χρήσης του άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας. Άρα λοιπόν η ανάγκη για τα project CCS είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το δουλεύουμε το θέμα, δεν μπορώ να σε υποσχεθώ τίποτα όμως για την ανακοίνωση. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλα έγγραφα υπό θέματα πιο μακροπρόθεσμα που αφορούν την ενέργεια και το κλίμα για μετά το 2020 και ίσως πρέπει να εντάξουμε και το CCS σε αυτή τη γενικότερη στρατηγική. Θα δούμε. Θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Αυτά είχα να πω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Chris Davis. Ευχαριστώ. Τι να πει κανεί. Είναι σε αυτή την κατάσταση. Σήμερα, με αυτή την τιμή του άνθρακα που έχει πέσει τόσο χαμηλά, τα πράγματα είναι σε τραυματική κατάσταση. Θέλω να φανταστούμε πάντως στη δεύτερη φάση ε, να υπάρξουν κάποια χρήματα και παρότι είναι ανοιχτό ο διαγωνισμό, υποτίθεται. Ε, τελικά η κρυψίνια είναι αυτή που κυριαρχεί. Από ό,τι φαίνεται μόνο ένας ενδιαφερόμενος ε, είναι. Μόνο η πρόταση της Ολλανδίας για το υδρογόνο φαίνεται να ε, ενδιαφέρεται για αυτό το διαγωνισμό. Είναι καλό να δει κανεί κάτι. Ε, τέλος πάντων, ένα project τουλάχιστον από το τίποτα καλύτερο είναι. Μακάρι να είχαμε περισσότερα. Και επανέρχομαι πάλι στις 100 χώρε. Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Υπάρχει κάποια ευελιξία για τα κονδύλια για να ξεπεράσει το πρόβλημα. Γιατί έχουν ήδη δοθεί χρήματα σε μια σειρά project στην Ευρώπη που τελικά δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστρέψουν στο γενικό προπολογισμό. Ή μάλλον πρέπει να είναι ακόμη στο γενικό προπολογισμό γιατί δεν έχουν δοθεί. Ρωτώ, υπάρχει μια κάποια ευελιξία εν προκειμένου για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα, για να φανώ και λίγο πιο αισιόδοξο. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχώ μου λέει ότι ε, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν με το CCS γιατί έχουν δώσει αρκετά κεφάλαια και πιστεύουν ότι υπάρχει ένας μηχανισμός παραγωγής εσόδων. Απλά εγώ δεν βλέπω στην πράξη να γίνεται τίποτα. Ούτε αποφάσει να λαμβάνονται εν ώψη των εκλογών που θα γίνουν σε δύο χρόνια. Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό στην ημερησία διάταξη. Ολοκληρώσαμε και το σύνολο της ημερησίας διάταξής μας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τη συνάδελφο και τον συνάδελφο που άντεξαν μέχρι το τέλος. 18-19 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίασή μας εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, από τις 3 μέχρι τις 6.30 την πρώτη μέρα και από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6.30 το βράδυ. Σας εύχομαι καλή επιστροφή. Καλό βράδυ. Λήξη της συνεδρίασης.